σας καλωσορίζω και εκ μέρους του συναδέλφου μου ε, Ζαν Αρτουή. Καλωσορίζω και τους δύο υποψηφίους ε, για τις θέσεις του Γενικού και τον Υπουργή Γενικού Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, τον κύριο Μόρτα και την κυρία Σιανόβα. Καλώς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως γνωρίζετε το άρθρο 7.6 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων ε, ορίζει τη διαδικασία με την οποία μέσω μιας ανοιχτής και διαφανούς ε, διαδικασίας ε, το Διοικητικό Συμβούλιο επιλέγει έναν υποψήφιο για κάθε μία από τις θέσεις ε, γενικού και αναπληρωτή γενικού διευθυντή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να ενημερώνονται έγκαιρα σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας επιλογής βάσει συγκεκριμένων ε, απαιτήσεων ε, εμπιστευτικότητας και αυστηρών απαιτήσεων. Έτσι λοιπόν ενημερωθήκαμε επίσημα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επιλέξει τον Βίλιαμ Μόλτερ και την Ιλιάνα Τσανόβα για τις δύο αυτές θέσεις. Και τώρα εδώ λοιπόν ε, θα λάβουν χώρα από κοινού οι δύο ακροάσεις και για τις δύο επιτροπές και θα ακολουθήσει η ψηφοφορία για τον διορισμό τους. Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με τη διαδικασία θα ξεκινήσουμε με μια εισαγωγική παρουσίαση. Ε, περνάμε τώρα στο βήμα της ακρόσης του William τα Θα μας παρουσιάσει τις αρχικές του σκέψεις για πέντε λεπτά και μετά υπάρχει δυνατότητα για τους συγητές και τους κοιόδης να υποβάλουν ερωτήσεις. Είναι φυσικά σημαντικό το βήμα αυτό, διότι το Κοινοβούλιο ε, συνέβαλε και είχε δεσμευτεί για την ταχεία υλοποίηση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Το Κοινοβούλιο επίσης ε, συνέβαλε στη βελτίωση της ποιότητας του κανονισμού και στο να κάνει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ένα μέσο που θα παράσχει και θα κινητοποιήσει επιπλέον επενδύσει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τώρα βρισκόμαστε στη φάση υλοποίηση και φυσικά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ισχυρή ομάδα ώστε οι δυνατότητες του EFSI να συναδούν με τις φιλοδοξίες και τις διατάξεις του κανονισμού στον οποίο συμβάλλουμε και εμείς ως συνομοθέτες. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε, ακόμα προσέρχονται οι συνάδελφοι, οπότε καθυστερώ λίγο για να μπει περισσότερος κόσμος στην αίθουσα, για να έχετε μεγαλύτερο ακροατήριο, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν κύριε Μόλτερ και πάλι καλώς ορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας κύριε και κύριοι. Με χαρά μου βρίσκομαι πάλι ενώπιόν σας ε, και υποψηφίου για το διορισμό του Γενικού Διευθυντή του ΕΦΣΥ. Να σας πω δύο λόγια για το παρελθόν μου. Για πολλά χρόνια ε, ήμουν ε, στο Αυστριακό Κοινοβούλιο, ήμουν υπεύθυνο για γεωργική πολιτική, για οικονομικά περιβαλλοντικά ζητήματα. Κατά τη διάρκεια της ε, χρηματοοικονομικής ε, κρίσης ε, κυρίως το 2007 και το 2008 και μέχρι πρόσφατα ήμουν ένας από τους αντιπροέδρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που είχαμε ως έργο μας μεταξύ άλλων και τις προκλήσεις της οικονομικής κρίσης. Προκλήσεις οι οποίες είναι τεράστιες Καταρχάς πρέπει οι Ευρωπαίοι πολίτες να βρουν θέσεις απασχόλησης. Είναι κάτι που πλήττει κυρίως τους νέους ανθρώπους που μαστίζονται από μεγάλη ανεργία. Έπειτα, να ενισχυθεί η βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης, να αυξηθεί μετά η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και γενικότερα της ευρωπαϊκής οικονομίας και να κλείσουν τα εφιστάμενα επενδυτικά κενά στην Ευρώπη. Επενδυτικά κενά τα οποία είναι τεράστια σε σχέση με το 2007. Αυτή είναι μια συστημική κρίση. Γι' αυτό αυτό που χρειάζεται είναι μια περιεκτική και ολοκληρωμένη πολιτική και αυτό το Ταμείο Στατικών Επενδύσεων είναι η απάντηση στη συστημική αυτή κρίση. Κυρίε και κύριοι, α μην ξεχνάμε ότι αυτό το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη αποτελείται από τρει πυλώνε και όλοι αυτοί διασυνδέονται και είναι εξίσου σημαντικοί. Καταρχά, πρέπει να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον φιλικό προς τις επενδύσεις και σε επίπεδο κρατών μελών και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να ολοκληρωθεί η ενιαία αγορά, η ενεργειακή αγορά, η ψηφιακή αγορά και να αρθούν τα εμπόδια και οι φραγμοί για τις επενδύσεις. Έπειτα, πρέπει να στηριχτούν οι επενδύσεις στην πραγματική οικονομία. Αυτό τι σημαίνει. Πρέπει να δημιουργηθεί καλύτερη στήριξη, καλύτερη ε, συμβουλευτική διαδικασία μέσω του European Advisory Hub και τρίτον να κινητοποιηθούν οι επενδύσεις, κάτι που θα βοηθήσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Κινητήρη μοχλή πίσω από αυτό θα είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά τη δεδομένη στιγμή. Δεν έχουμε πρόβλημα ρευστότητα στην αγορά. Υπάρχει ρευστότητα στην αγορά. Τα προβλήματα υπάρχουν από τη μία στην ε, περιορισμένη δυνατότητα ανάληψης κινδύνου των εμπορικών τραπεζών και στην ε, υποανάπτυκτη κεφαλαία αγορά που έχουμε στην Ευρώπη. Υπάρχει νομοθεσία που προβλέπει αυτή την ε, εγγύηση 21 δισεκατομμυρίων που θα δώσει τη δυνατότητα στο ΕΕΦ να αυξήσει τη δυνατότητα αντιμετώπισης κινδύνου και να δώσει τη δυνατότητα λοιπόν για επενδύσεις στην πραγματική οικονομία. Αυτό που έχουν καταφέρει οι βουλευτές ε, των Ηνωμένων Πολιτειών με τον κανονισμό ΕΦΣΑ είναι ότι καταρχάς αυτά τα 21 δισεκατομμύρια στηρίζουν και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 5 δισεκατομμύρια ευρώ ε, και έπειτα την ύπαρξη αυτού του πυλώνα υποδομών που στηρίζεται από 16 δισεκατομμύρια ο οποίος θα στηριχθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Επίσης, έχετε ακούσει όλοι για την περαιτέρω κινητοποίηση 350 δισεκατομμυρίων ευρώ τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει ένα πλαίσιο λοιπόν που μας προσφέρει σαφείς κανόνες και σαφή καθοδήγηση και σαφείς στόχους. Να σας υπενθυμίσω ότι το άρθρο 5, το οποίο μας δίνει συγκεκριμένες ενδείξεις για το τι σημαίνει additionality, Υπάρχουν κριτήρια επιλεξιμότητας, αναφέρεται το τι χρειάζεται για να επιτευχθεί αυτή, αυτός ο στόχος. Μετά αναφέρονται οι γενικότεροι στόχοι στο άρθρο 10. Δημιουργείται μια σαφή εικόνα των μέσων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να επιτεύξουμε το στόχο αυτό. Και ο κανονισμός αυτός θα δώσει μια νέα ευκαιρία Μέσω της συνεργασίας με τις εθνικές τράπεζες, με τις εθνικές επενδυτικές πλατφόρμες και θα παρέχει επίσης στήριξη σε διασυνοριακά προγράμματα, τα οποία είναι απολύτως αναγκαία, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για έργα υποδομών. Επίσης, μας δίνει έναν ξεκάθαρο προσανατολισμό για τις επενδύσεις ε, και καθοδηγεί το εποπτικό όργανο του ΕΦΣΥ. Αυτό θα δοθεί μέσω του δίκτυου επιδόσεων, για παράδειγμα, και μέσω της, ε, των καθετευθυντηρίων γραμμών για την ε, βιωσιμότητα. Το, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχουν στο ταμείο αυτό, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το European Advisory Hub θα συντίθεται λοιπόν από εκπροσώπους όλων των θεσμικών οργάνων. Ο κανονισμός ΕΦΣΑ λοιπόν μας δίνει έναν ξεκάθαρο προσανατολισμό και ξεκάθαρες εγκατευθυντήριες γραμμές για τον γενικό του διευθυντή και το διοικητικό συμβούλιο. Ο γενικό διευθυντής είναι υπεύθυνο για τι καθημερινέ εργασίε, ο εκτελεστικό διευθυντής είναι υπεύθυνο για την διοίκηση και την λήψη αποφάσεων στι επιμέρου επιτροπέ και επίση είναι αρμόδιο έτσι ώστε να γίνεται η καλύτερη δυνατή προετοιμασία ε, το, της υποβολής εκθέσεων. Και υπεύθυνο για τις ε, σχέσεις με τις ε, εθνικές τράπεζες, με τα εθνικά ιδρύματα, το European Advisory Hub και τα υπόλοιπα συμμετέχοντα όργανα. Αυτό είναι το κεκτημένο λοιπόν που μας δίνει ο κανονισμός. Συντονισμός με τις διάφορες υπηρεσίες με το Investment Hub και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έπειτα, μαζί με την ΕΤΕ θα εντοπίσουμε τους κοινού στόχους με τις Εθνικές Τράπεζες, κοινά διασυνοριακά έργα, θα στηριχτεί η ανάπτυξη καινούριων έργων βασισμένα στα ήδη ε, υφιστάμενα έργα, μικροχρηματοδότηση για παράδειγμα, επενδύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσει, και επίση να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει μια κοινή άσκηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΤΕ έτσι ώστε να ε, γίνει το ε, γνωστό όχι μόνο στους ε, δημόσιου επενδυτέ, αλλά κυρίω στους ιδιωτικού φορεί που θα επενδύσουν. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό ευθύ εξ αρχή να τεθούν οι κανόνε για την υποβολή εκθέσεων και για του ελέγχου και είναι πάρα πολύ σημαντικό οι συντονιστέ να είναι σε συνεχή επαφή με του ε, εμπλεκόμενου φορεί. Ένα από του οποίου είναι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χρειάζονται, χρειάζεται βελτίωση, χρειάζεται βελτίωση επιγόντως, διότι είναι προς το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών να ολοκληρωθεί η διαδικασία το ταχύτερο δυνατόν. Το, ο κανονισμός ΕΦΣΑ δεν είναι το μαγικό ε, ραβδί, όμως είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στατικό στοιχείο των ε, σημαντικών πυλώνων για την Ευρώπη. Και η δική μου υποχρέωση και δικός μου στόχος και η πεποίθηση που έχω είναι ότι ο ΕΦΣΑ είναι ένας από τους ε, βασικούς ε, τρόπους που μπορούμε να στηρίξουμε τον ευρωπαϊκό τρόπο σκέψης. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας που με άκουσε και σας καλώ μαζί να κάνουμε το ΕΦΣΙ επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα δίνουμε το λόγο στον Χωσέ Μανώλη Φερνάντα για την πρώτη ερώτηση. Δύο λεπτά έχετε στη διάθεσή σα. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να καλωσορίσω και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών, τον εισηγητή Πούλμαν και τους υποψηφίους. Στρέφομαι στον κύριο Μόλτερερ καταρχάς διατελέσατε μέλος ε, του Διοικητικού Συμβουλίου της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και είχατε τη θέση του Αντιπροέδρου. Φαντάζομαι ότι αυτό σας έχει δώσει σημαντική εμπειρία, η οποία θα σας φανεί χρήσιμη και για τις στρατηγικές <laughs> επενδύσεις, για το Ευρωπαϊκό τέμιο Στρατηγικών Επενδύσεων, αλλά ενδεχομένως από την άλλη πλευρά να έχουμε ένα θέμα ε, με την έννοια της προσθετικότητας. Το Κοινοβούλιο δεν επιθυμεί το ΕΦΣΙ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατικών Επενδύσεων, να επαναλάβει ή να επικαλύπτει άλλους οργανισμούς. Πώς θα εγγυηθείτε λοιπόν και την πλήρη ανεξαρτησία, ε, επιχειρησιακή και λειτουργική ανεξαρτησία ταμείου. Απάντηση. Είναι σαφής ο κανονισμός. Το μόνο καθήκον του ε, διευθυντή είναι να λειτουργεί το ΕΦΣΙ σωστά και να τηρεί πλήρως τις διατάξεις του κανονισμού. Τελεία. Έπειτα έχουμε οκτώ ανεξάρτητα μέλη που απαρτίζουν την Επιτροπή Επενδύσεων. Η Επιτροπή Επενδύσεων είναι ο μόνος φορέας που θα αποφασίσει για την επικύρωση των εγγύσεων τρίτων. Πιστεύω ότι η συμμετοχή στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό εθνικών τραπεζών προώθησης αλλά και ιδιωτικού κεφαλαίου θα δώσει αυτή τη νέα όθηση που είναι και απολύτως αναγκαία και θα υπάρχει ε, αυτή η προσθετικότητα. Γιατί αυτή είναι η έννοια της προσθετικότητας. Ε, έχουμε ένα ε, προφίλ πιο υψηλού κινδύνου, ειδικό κεφά, ιδιωτικό κεφάλαιο που συμμετέχει σε επενδύσεις, κατά δεύτερον και κατά τρίτον το συμβουλευτικό κομμάτι, η συμβουλευτική συνιστόσα. Και υπάρχει και μια τέταρτη συνιστόσα, όπω είπα και στην εισαγωγή μου, που είναι η ανάπτυξη νέων προϊόντων αλλά επαναλαμβάνω ότι εγώ δεσμεύομαι ότι θα τηρώ τον ε, κανονισμό, τον πούλμα. Ε, Κύριε Μόλτερε, σήμερα το πρωί συναντήθηκα με τον πρόεδρο της ΕΤΕ, τον κύριο Μάλιστατ, ε, σε ένα πάνελ που συζητούσαμε τα επιτεύγματα του κανονισμού ΕΦΣΥ και άνοιξε λοιπόν την ομιλία του λέγοντας ότι αφού του είδε ότι έγινε Ό,τι έκανε συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αυτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέκτησε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από πριν. Έγιναν πολλές αλλαγές στο αρχικό σχέδιο, στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μας είπατε και εσείς για τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις κατευθυντήριες γραμμές για τις επενδύσεις, τον πίνακα επιδόσεων. Όλα αυτά όμως επετέφθησαν ας το πω έτσι, παρά τους δισταγμούς που είχαν διατυπωθεί. Από τη μία της ΕΤΕ και από την άλλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έπρεπε λοιπόν να το παλέψουν τον κανονισμό αυτό. Υπάρχει μια τάση, ο κανονισμός εύση, αντί να θεωρείται ένα νέο μέσο, να θεωρείται ένας ε, ξεχωριστός λογαριασμό ε, μέσα στα, στην ε, ΕΤΕ. Εσείς πώς θεωρείτε ε, ότι θα μας πείσετε πως αυτό είναι κάτι νέο ως εκπρόσωπος του παλιού, των παλιών δομών. Αυτή είναι, αυτό είναι αποφασιστική σημασία για εμένα. Καταρχάς, κύριε Μπούλμαν, Είστε έμπειρος πολιτικός και δεν θα σας ε, εκπλήσει το γεγονός ότι σε μια διαπραγμάτευση πρέπει να ξεπεράσετε εμπόδια. Αυτό συμβαίνει στην ε, πολιτική. Ναι, ε, οπότε λοιπόν μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι έχουν γίνει πολλά. Εν συγκρίνουμε την αρχική πρόταση του κανονισμού με το τελικό αποτέλεσμα, βλέπουμε ότι έχουν επιτευχθεί πολύ σημαντικά πράγματα και από εσά. Οι, οι γραμμέ για την εταιρική επενδυτική πολιτική, για παράδειγμα, δεν το αρνούμε αυτό. Εσείς αυτό που καταφέρετε να εισαγάγετε ε, σχετικά με την υποβολή εκθέσεων και με τους ελέγχους είναι πάρα πολύ σημαντικό και τονίζει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο πυρήνας της δημοκρατίας. Δεν ήμουν υπάλληλο στην ΕΤΕ, διορίστηκα για τέσσερα χρόνια στο, στην δίκηση της ε, τράπεζας και ως μέλος της ε, δικού σας επιτροπής απέκτησα μια καλή εικόνα για το τι πρέπει να αλλάξει. Και πιστεύω πως το ΕΦΣ είναι ένα όργανο το οποίο μας προσφέρει πολλά περισσότερα από τα εφιστάμενα. Μας δίνει νέου ε, νέους τρόπους να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε ενωπιών μας. Και εσείς ως θεματοφύλακες των συνθήκων έχετε ως καθήκον να, να προσέξετε να εφαρμοστεί αυτός ο κανονισμός. Ο Γενικός Διευθυντής λοιπόν είναι αρμόδιος μόνο για το ΕΦΣΥ. Τελεία. Για τίποτα άλλο. Και να είστε σίγουρος ότι οι εμπειρογνώμονες της ε, Επιτροπής ξέρουν πολύ καλά τι ε, περιέχει ο κανονισμός και ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές της επενδυτικής πολιτικής. Ξέρουν αυτές τις λεπτομέρειες. Έχετε μια ερώτηση ως συνέχιση αυτής. Όχι. Ξεκινάμε με τους ε, σκιώδεις εισηγητές των δύο ε, επιτροπών για το ΕΛΚΟ Ατμαρκάρας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μόλτερερ, το ερώτημα παραμένει το ίδιο. Θέλουμε ένα εύση που δεν θα είναι ένα αυτόματο μηχάνημα ανάληψης μετρητών της ΕΤΕ. Θέλουμε ανεξαρτησία από τη μία και από την άλλη θέλουμε ορισμέ... εγγυήσεις για την ε, προσθετικότητα. Γι' αυτό λοιπόν σας ερωτώ ξανά, ποια βήματα θα κάνετε εσείς ως γενικός διευθυντής έτσι ώστε να διασφαλιστεί αυτή η προσθετικότητα και να αποφευθούν τα οι συνήθεις πρακτικές. Ε, έπειτα, ποιες θα είναι οι προκλήσεις, οι ρυθμιστικές, νομοθετικές, πολιτικές, οικονομικές ε, στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ΕΦΣΥ και ποια στρατηγική θα υιοθετήσετε για να τις αντιμετωπίσετε. Και τρίτον, τα χρήματα για τα έργα που θα υπαχθούν στο ΕΦΣΥ, από πού θα έρθουν, από ιδιωτικού φορείς και αν από ιδιωτικούς φορείς εσείς πώς θα διασφαλίσετε ως γενικός διευθυντής ότι τα έργα αυτά θα καταναμηθούν δίκαια σε όλα τα κράτη-μέλη και δεν θα επικεντρωθούν σε λίγα από αυτά έτσι ώστε να πάει και η πλειοψηφία των κονδυλίων σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Η απάντηση. Δύο ερωτήσεις θα γίνουν από κοινού. Ο κύριος αν έχει το λόγο. Μετά θα απαντήσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τρία σχόλια από πλευρά μου. Πρώτα απ' όλα, κύριε Μόλτερ, πώ θα προλάβετε ανομοιόμορφη γεωγραφική κατανομή των έργων, ακόμη και στην περίπτωση όπου η μεγάλη πλειοψηφία των επιλέξιμων έργων θα προέρχονται από μικρά πολυάριθμα κράτη-μέλη και από συγκεκριμένε περιοχέ τη Ευρώπη. Και εδώ φυσικά πρέπει να λάβουμε υπόψη χώρες με λιγότερα ανεπτυγμένες ε, χρηματοπιστωτικές αγορές που έχουν ελάχιστη εμπειρία με τέτοιου είδου χρηματοπιστωτικά μέσα. Δεύτερη, όσον αφορά τον κόμβο, πώς βλέπετε τη συνεργασία με τις εθνικές και ειδικότερα με τις περιφερειακές αρχές ε, ώστε να διασφαλιστεί ευρύτερη πρόσβαση σε πιθανούς δικαιούχους βοήθειας από τον κόμβο. Και τρίτον, ε, για το γενικό σας ρόλο ως Διευθυντού Συμβούλου σκοπεύετε να ασκήσετε το ρόλο αυτό ως Διευκολυντής ε, για περιφερειακές αποφάσεις εντός της ε, Επιτροπής ή σκοπεύετε να εμπλακείτε ενεργά δεδομένου ότι η Επιτροπή σας λαμβάνει αποφάσεις με απλή πλειοψηφία από όσο γνωρίζω. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. πρώτα απ' όλα για τον κύριο Κάρας για μένα κλειδί του FC είναι ότι παρέχει αυτή την προσθετικότητα όπως περιγράφεται στον κανονισμό σε συνδυασμό με την επιλεξιμότητα όπως επίσης περιγράφεται στον κανονισμό αυτό σημαίνει αντιμετώπιση ε, προβλημάτων των αγορών αγράφεται στον κανονισμό αυτό δεύτερον να γίνουν επενδύσεις δυνατές οι οποίες δεν είναι δυνατές χωρίς το ΕΦΣΕ υψηλότερο προφίλ κινδύνου σε σχέση με το σημερινό προφίλ κινδύνου της ΕΤΕ, κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και τεχνικά και οικονομικά βιώσιμα έργα. Αυτά είναι τα κριτήρια, τα οποία μάλιστα αποτελούν ε, βάση και για το πίνακα αποτελεσμάτων, το scoreboard που διαπραγματευτήκατε και για τις αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου για να επιτευχθεί ο πολλαπλασιαστής που αποτελεί και αυτός κομμάτι της συζήτησης και για το κοινό είναι σαφές ότι αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να πληρούνται διότι διαφορετικά είναι δύσκολο να υπάρξει ο πολλαπλασιαστής είναι πώς μας φέρει όλους να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Δεύτερον, κλειδί για τα πρώτα δύο-τρία χρόνια είναι ανάπτυξη έργων, ανάπτυξη έργων, ανάπτυξη έργων. Διότι αυτό που μας λείπει ό,τι θα μας λείπει στην πρώτη περίοδο θα αντιστοιχεί σε έλλειψη πραγματικών επενδύσεων της δεύτερης περίοδου. Οπότε ανάπτυξη έργων, αυτό χρειάζεται. Και τρίτον, όσον αφορά τους όρους για την περιφερειακή κατανομή. Νομίζω ότι στην ε, κατευθύντρια γραμμή ε, αναφέρεται σαφώς ότι πρέπει να αποφύγουμε συγκέντρωση σε συγκεκριμένους τομείς ή σε συγκεκριμένες χώρες. Αυτό πρέπει να είναι είναι ότι το ΕΦΣΙ δεν θα είναι το ίδιο για όλες τις χώρες. Για να υπάρχει ευελιξία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Τέσσερις χώρες με εθνικές ε, τράπεζες προώθησης και ε, άλλες χώρες με ιδρύματα αντίστοιχα προώθησης και άλλες χώρες που ενδιαφέρονται να προετοιμάσουν ε, πλατφόρμες, άλλες είναι έτοιμες για διασυνοριακές συναλλαγές και αυτή πρέπει να είναι η ευελιξία μας ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες των αγορών που διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Και η περιφερειακή κατανομή θα ε, υποστηριχθεί από το κέντρο επενδύσεων. Αυτό είναι ε, το κλειδί. Το Συμβουλευτικό Κέντρο Επενδύσεων είναι έτοιμο να υπογράψει σύντομα ένα μνημόνιο συνεννόησης με τους ε, εταίρους στα κράτη-μέλη και φυσικά στη συνέχεια να διευκολύνει με αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη επενδύσεων. Εγώ δεν είμαι διευκολυντής. Θα δράσω προενεργά ώστε να γίνει δουλειά. Ευχαριστούμε. Θέλω να παρακαλέσω τους συναδέλφους ε, να μην υπερβαίνουν το 1,5 λεπτό στις ερωτήσεις τους ώστε να έχουμε και αρκετό χρόνο και 1,5 λεπτό θα είναι και η απάντηση. Η Έιντερ Γκαρθιατάμπαλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μόρτερε. Είχα δύο πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις ε, στην εισαγωγή σας. Μιλήσατε για το ότι αυτή η Επιτροπή Επενδύσεων πρέπει να είναι ανεξάρτητη σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις που θα πρέπει να λαμβάνει. Θα ήθελα να μου πείτε όμως εσείς πώς βλέπετε τη σχέση που θα πρέπει να έχετε εσείς με την Επιτροπή Επενδύσεων για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει αλληλεπικάλυψη καθηκόντων ούτε θα παραμένουν κάποιοι τομείς ακάλυπτοι. Δεύτερο ερώτημα, είπατε ότι ο στόχος σας ο απότατος ουσιαστικά είναι να λειτουργήσει αυτό το ταμείο να ολοκληρωθεί, να είναι επιχειρησιακό, να πετύχει τους στόχους του. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που μου έχουν γνωστοποιήσει πολλές επιχειρήσεις είναι ότι δεν γνωρίζουν πώς να απευθυνθούν στο Ταμείο. Φαντάζομαι ότι και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα το ίδιο συνέβαινε και δεν σας ε, πρόξενει έκπληξη αυτό. Πώς εσείς θα βοηθήσετε οι επιχειρήσεις και οι δύο συγκρομεσίες επιχειρήσεις να μπορούν πραγματικά να συμμετέχουν στο Ταμείο αυτό. Ευχαριστώ. Η Ελίζα Φερέιρα τώρα. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Είπατε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι θεματοφύλακας, ε, ένας από τους θεματοφύλακες. Μέχρι τώρα όμως δεν καταφέραμε να έχουμε μια διοργανική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, άρα αυτό γύρει ένα ζήτημα. Και ρωτώ, εσείς αν επιβεβαιωθείτε σε, σε αυτή τη θέση, σε αυτό το αξίωμα, ε, θα φροντίσετε να έχουμε ε, μια διοργανική συμφωνία όπως έχουμε ε, με την ΕΚΤ για παράδειγμα ε, για την πλήση διαφορά των σχετικών μηχανισμών κτλ. Δεύτερο ερώτημα. Μέχρι τώρα δεν είχαμε τη δυνατότητα να είμαστε ένα σταματοφύλακα να ελέγχουμε το τι γίνεται και αν δεν υπάρξει η διοργανική συμφωνία ο αριθμό 6 του κειμένου που λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ότι τηρούνται ενήμερα με το δέοντα και έγκαιρο τρόπο για όλα τα στάδια τη διαδικασία επιλογή για αυτό το αξίωμα. Αφού δεν πήραμε όμως καμία πληροφορία, εσείς είστε, όπως είπατε, στη διεύθυνση, στη διοίκηση, λοιπόν, που τα λέω έτσι ομάλα, δεν είναι ξεκάθαρο. Αν υπάρχουν σαφείς σε περιπτώσεις σύγκρουση συμφερόντων, τι γίνεται. Αν προτείνει η διοίκηση έναν και μόνο υποψήφιο και εμείς πρέπει να τον εγκρίνουμε. Επίσης, να κάνω και ένα άλλο ερώτημα σε σχέση και με το καταστατικό της ΕΤΕ υπάρχει το πρωτόκολλο υπαρθμών 28 για την οικονομική, κοινωνική και δαφική συνοχή. αμφιβάλλω ότι η ΕΤΕ τήρησε αυτή την εντολή. Τι διαφορά ε, θα έχει το Ταμείο όταν θα έχει μια παρόμοια εντολή για το αξίωμα αυτό. Και εσείς συγκεκριμένο ο κύριος Μόρτερ για να απαντήσει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ο αναφέρει σαφώς ότι ο Διευθύνων Συμβουλός προεδρεύει το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Γενικός Διευθυντής. Αυτό γράφεται και στο κανονισμό ψηφίζει, στη Διοικητικό Συμβούλιο και μαζί με τον αναπληρωτή προετοιμάζει την Επιτροπή Ερευνών, δίνει τις σχετικές εντολές για τις για τις επενδύσεις, ε, συγγνώμη, και της Επιτροπής Επενδύσεων, με σκοπό όχι να καθυστερεί τη διαδικασία αλλά να επικυρώνει την διαδικασία λήψης αποφάσεων. Δεύτερον, πώς προσεγγίζουμε το ΕΦΣΙ, υπάρχουν πολλές επιλογές μέσω της ΕΤΕ, μέσω των Εθνικών ε, Ιδρυμάτων Πρόθεσης και αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι το Συμβουλευτικό Κέντρο Επενδύσεων είναι ήδη ένα σημείο εισόδου επαφής με, με το ΕΦΣΙ. Αυτό το γνωρίζω από συναδέλφους. Και Βέβαια, όπως είπα, θα υπάρξει αυτή η άσκηση πρόθεση κάτι πρέπει να κάνουμε από κοινού μαζί με την ΕΤΕ, ώστε να γίνει αυτό δυνατόν και να το γνωρίσουμε στον τραπεζικό τομέα. Τώρα, όσον αφορά τη συμφωνία, η διαπραγμάτευση με το Κοινοβούλιο και την ΕΤΕ συνεχίζει ε, για τη συμφωνία εμπιστευτικότητας. Βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις, στις οποίες εγώ δεν συμμετέχω. Για να διευκρινίσω, υπήρξα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Όταν δημοσιεύτηκε η θέση, αμέσως ρώτησα την Επιτροπή Ηθικής και Συμμορφωσής μας και είπα τι πρέπει να κάνω για να ε, ε, κάνω αίτηση για αυτή τη θέση και πληρούσα ακριβώς όλες τις απαιτήσεις της Επιτροπής Ηθικής και Συμμόρφωσης της ΕΤΕ. Φυσικά μετά από την αίτησή μου δεν, υπήρξα, δεν συμμετείχα σε καμία απόφαση. Απήχα από οποιοδήποτε είδους απόφαση της ΕΤΕ. Και αυτό είναι απόλυτα σαφές. Τρίτον, η ΕΤΕ ασχολείται με πολλές εντολές για επιχειρήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την καινοτομία και σε συνεργασία με το RSFF. Η διαχείριση εντολών είναι συνήθεις εργασίες ε, της ε, ΕΤΕ. Εδώ μιλάμε για μια πρόσθετη εντολή, με πολύ σαφείς ε, γραμμές. Δεν είναι κάτι καινούριο, είναι επιπλέον, είναι συμπληρωματικό και δεν έρχεται σε αντίθεση με τη συνοχή. Πιστεύω ότι το ΕΦΣΙ συμπληρώνει την πολιτική συνοχής. Ευχαριστούμε. Ας περάσουμε στην ομάδα ECR. Ο κύριος Άσκροφτ. Όχι. Σανδολούνας. Έχει και άλλους ομιλητές στο ECR που θέλουν να λάβουν το λόγο. Δεν είναι υποχρεωτικό φυσικά. Okay, so we go to the ALDE group. Λοιπόν, εκ μέρους του, ε, ε, του ALDE ο κύριος Νίλ Στορβάλ, όχι, ο κύριος Τρεμόσα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις ε, εντός ενός λεπτού. Στις συζητήσεις για το ΕΦΣΥ είχαμε δύο προτεραιότητες. Η μία από αυτές τελικά καταφέραμε να γίνει η ανάλυση κόστους ωφέλους για να δούμε τη διαδικασία ορισμένα κράτη-μέλη ή υπεράσπισαν το να κρατήσουμε το status και να υπάρξουν εθνικές αναλύσεις ωφέλους, Οπότε θα υπάρξει πίεση να, για να συνεχιστούν οι επενδύσεις ε, σε έργα που ενδεχομένως να μην είναι τα καλύτερα για την ευρωπαϊκή οικονομία. Πώς θα αντισταθείτε σε αυτή την πίεση των κρατών μελών. Δεύτερο, στο τελικό κείμενο καταφέραμε να δώσουμε κάποια προτεραιότητα στα ευρωπαϊκά δίκτυα ε, και στα σχετικά επενδυτικά έργα όσον αφορά την ενέργεια και τις μεταφορές. Κάτι που συζητήθηκε εδώ, συζητείται εδώ και τα τελευταία πέντε χρόνια σε αυτό το κοινοβούλιο. Μάλιστα σε ορισμένα κράτη-μέλη δεν υπάρχει καμία διασύνη επένδυση ή χρηματοδότηση τέτοιων εργών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώ εσεί λοιπόν θα δώσετε όθηση σε τέτοια έργα. Ο κύριος Ντεπρέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απευθύνομαι στους ε, υποψηφίους. Διάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον ε, το βιογραφικό σας ε, που μας δώσατε και έχω δύο παρατηρήσεις. Ήσασταν ένας επαγγελματίας που από τα 35 χρόνια, με 25 χρόνια, στα 25 χρόνια ασχοληθήκατε με τη γεωργία. Ήσασταν άνθρωπος λοιπόν ενός τομέα. Και μετά κοιτάω παραπέρα και έχετε καμιά δεκαριά χρόνια που ανήκατε σε ένα κόμμα. Λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι δεν γνωρίζω τίποτα. Είμαι ένας απλός πολίτης και διαρωτώ με ο άνθρωπος αυτός που έκανε ένα επάγγελμα και μετά ανήκε σε ένα κόμμα τι εγγύσεις μπορεί να προσφέρει, πώς εμφανίζεται μπροστά μου και προσπαθεί να με κάνει να πιστέψω ότι θα ε, εφαρμόσει όσα προβλέπονται στο καταστατικά. Ε, και έχω και μια πιο συγκεκριμένη ερώτηση. Στο άρθρο 7 παράγραφος 9 αναφέρεται ότι ο πρόεδρος πρέπει να επιβλέπει ώστε η Επιτροπή Επενδύσεων να λαμβάνει αυτόνομα τις αποφάσεις της και επίσης προβλέπεται οι οργανωτικές διευθετήσεις να καθορίζονται και να διατηρούνται ώστε να λειτουργεί σωστά η Επενδυτική Επιτροπή. Μπορείτε να μου πείτε πώς προβλέπετε να γίνεται η οργάνωση αυτής της ε, οργανωτικής αυτονομίας. Ευχαριστώ κύριε Μότερα. Πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η σχέση κόστους όφελους. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει και ο δείκτης επιδόσεων και οι μετρήσεις που βασίζονται σε αυτόν. Είναι μια σαφής ένδειξη για την Επενδυτική Επιτροπή της ώστε να μπορέσει να λάβει αποφάσεις. Επαναλαμβάνω, η ε, Επιτροπή Επενδύσεων αποτελείται από ε, οκτώ ανεξάρτητα μέλη, όχι κράτη-μέλη. Είναι η... το Διοικητικό Συμβούλιο που ε, ασκεί τα καθήκοντά του βασισμένο στον κανονισμό, στο καταστατικό. Και είμαι σίγουρος πως ξέρετε απολύτως ε, τι είναι το σημαντικό και εδώ είναι η ευρωπαϊκή διάσταση. Έπειτα, το δίκτυο και οι υποδομές. Πιστεύω πως είναι τα βασικότερα ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθεί το ΕΦΣΙ και αυτά που παρατηρώ από την αγορά είναι ότι υπάρχει μια ζήτηση για ενεργειακό δίκτυο, για κλασικές υποδομές, για νέες ε, υποδομές και εδώ έρχονται και οι πρωτοβουλίες ε, που θέλουμε να λάβουμε και για διασυνοριακά έργα. Και ο Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής μάλιστα έχει τοποθετηθεί σχετικά. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία είναι τα βασικότερα ε, στοιχεία των δραστηριοτήτων μας. Έπειτα, πράγματι, προέρχομαι από το χώρο της Γεωργίας και είμαι περήφανος γι' αυτό. Καταρτίστηκα στην Γεωργία, υπηρέτησα ως υπουργό Γεωργίας, όμως ε, το ότι ήμουν υπουργό Γεωργίας ε, δεν σημαίνει πως είμαι ε, αρμόδιος μόνο για τους αγρότες και εκπροσωπώ μόνο εκείνους. Οι αυστριακοί βουλευτές ξέρουν πολύ καλά πως η εντολή που έχω πρέπει να υπηρετεί τους πολίτες και η Γεωργία είναι μέρος της οικονομίας που υπηρετεί τους πολίτες. Και η εμπειρία μου τα τελευταία χρόνια, για να είμαι ειλικρινής, έχει δείξει ότι υπάρχουν τομείς όπου η πολιτική μπορεί να αλλάξει πράγματα. Υπάρχουν όμως και άλλοι τομείς στους οποίους η πολιτική δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το ΕΦΣΙ είναι ένας από αυτούς. Η ουσία μετράει εδώ. Δεν κρύβω απολύτως τίποτα. Πράγματι, ε, προέρχομαι από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, από συγκεκριμένο ε, χώρο, το χώρο της γεωργίας, ανήκω σε ένα συγκεκριμένο κόμμα. Τώρα όμως έχω φτάσει σε ένα διαφορετικό στάδιο της ζωής μου με διαφορετικές ευθύνες. Έχω κλείσει ένα κεφάλαιο και άνοιξε ένα άλλο. Και αυτό πιστεύω πως θα έπρεπε να είναι δυνατό και για έναν πολιτικό. Με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος. κύριος Μόλτερ Αναφερθήκατε και στην ΕΤΕ και το άρθρο 9. Θα, θα επανέλθω, εντάξει, μακρηγόρησα στα τελικά μου σχόλια. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρου τη ΓΚΟΕ τώρα, ο κύριος Φάμπιο Ντεμάζη. Καλησπέρα κύριε Μόλτερερ. Σε ορισμένες συνεντεύξεις σας ε, πρόσφατα μας είπατε πως ε, η Συμβάσει σε ιδιωτικού τομέα είναι πάρα πολύ σημαντικέ για να δώσουν όθηση στις επενδύσεις. Δεδομένης της ε, άσχημη κατάσταση των δημόσιων οικονομικών στα ορισμένα κράτη-μέλη και τον οποιονδήποτε λόγο, υπάρχουν προβλήματα χρηματοδότηση επενδύσεων μέσω αυτών των εταιρικών σχέσεων δημόσιου τομέα. Όμω, το γερμανικό ελεκτικό συνέδριο απεφάνθη ότι κοστίζει πάρα πολύ στον ε, φορολογούμενο Ε, αυτή, η επένδυση. Εσείς τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Έπειτα θα ήθελα να σας ρωτήσω για τα έργα τα οποία έχουν τρομολογηθεί μέχρι τώρα. Δεν έχουμε ακόμα τελειώσει τον τριμερή διάλογο. Γι' αυτό θα ήθελα να μάθω εσείς Πού βλέπετε το επίπεδο των επενδύσεων, ε, πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση και ποιες ε, είναι οι αποφάσεις που ε, έχετε κληθεί ως τώρα να πάρετε. Ποιες είναι οι τάσεις που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν τάσεις αντικατάστασης των δημόσιων επενδύσεων με αυτές τις επενδύσεις που θα προέρθουν από το ΕΦΣΥ. Υπάρχουν άλλοι ομιλητές από την ΚΟΕ, αν όχι να απαντήσετε κύριε Μόλτερ για τις ε, συμπράξεις ιδιωτικού τομέα. Είναι ένα ενδεχόμενο αυτό. Να έχουμε διαρθρωμένη χρηματοδότηση και αυτή είναι μία από τις δυνατότητες. Αλλά αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να αποφύγουμε είναι να έχουμε μία συζήτηση άσπρο ή μαύρο. Υπάρχουν σδίτη που λειτουργούν πολύ καλά και υπάρχουν σδίτη που δεν λειτουργούν πολύ απλά. Και αυτή είναι η προσέγγιση που θέλω να ακολουθήσω. Θέλω να βρίσκω την καλύτερη λύση. Αλλά αν θέλουμε το Ταμείο πραγματικά να γίνει πραγματικότητα, να προσελκύει ιδιωτικό κεφάλαιο δηλαδή, θα πρέπει, τα δείτε, αυτό το μοντέλο να χρησιμοποιηθεί ναι, ένα από τα μοντέλα για την προσέλκυση του ιδιωτικού κεφαλαίου. Ιδίω στη Γερμανία το γνωρίζω γιατί ε, ήμουν αρμόδιος για τις επιχειρήσεις στη Γερμανία κατά το παρελθόν ε, και αυτή η συζήτηση πραγματικά επηρεάζει και τη νέα δομή ε, των ΣΔΙΤΑ που προτείνει η γερμανική κυβέρνηση σήμερα. Αυτή είναι μια επιλογή. Το θέμα είναι ποια είναι η καλύτερη επιλογή. Αν είναι καλύτερη αυτή η επιλογή, καλώς. Αν όχι, επιλέγουμε κάτι διαφορετικό. Δεύτερον, αποθήκευση, warehousing. Από ό,τι κατάλαβα, ε, έχει ξεκινήσει, έχει, έχει δρομολογηθεί, Πρέπει πρώτα να συγκροτηθεί και να αρχίσει ε, να ασκεί τα καθήκοντά της η Επιτροπή Παιδείας. Η Κομισιόν ε, επικυρώνει την ε, εγγύηση και έπειτα γιατί προτείνει, παραδείγματος χάρη, ενέργεια. Είναι ένας από αυτούς του τομείς η ενεργειακή απόδοση, η καινοτομία, η κοινωνική κατοικία. Πολύ ενδιαφέρον τομέας. Μπορεί να επηρεάσει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές επιλύσεις και της προσφυγικής κρίσης. Σας δίνω απλά μια ιδέα για ορισμένα τέτοια παραδείγματα. Προείπα όμως και στον ε, κύριο Κάρας ότι θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε τις προσπάθειες εκπόνησης έργων. Είναι ένα από τα σημεία που πρέπει να αναπτύξουμε. Η δημόσια και ιδιωτικά έργα. Αυτός ο κατάλογος ε, των έργων του Δεκεμβρίου του 2014 ήταν ενδεικτικός. Κατέδειξε όμως σαφώς και πού υπολοιπόμεθα ακόμη, και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Έρνεστ Μαραγκάλ, εκ μέρους των Πρασίνων. Θέλετε το λόγο? Όχι. Κυρία Βάνα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Μόλτερ, ε, πριν το καλοκαίρι είχα ήδη τη δυνατότητα να, ε, στα πλαίσια της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης να σας υποβάλω ερωτήσεις για την διασφάλιση των κοινωνικών επενδύσεων στα πλαίσια του ΕΦΣΥ και να σας υποβάλω ερωτήσεις για την ποιότητα των στόχων και της δέσμευσης του ΕΦΣΥ στο Ευρώπη 2020. Μπορείτε εσείς τώρα στα πλαίσια της αίτησης ε, αυτής για Διευθυνόν Σύμβουλο του ΕΦΣΙ να, μας, ε, να μου απαντήσετε για το ποια νομίζετε πως θα είναι η συμβολή για τις ε, επενδύσεις που σχεδιάζονται έτσι ώστε να στηρίξουν πραγματικά την προσπάθεια που κάνουμε για το περιβάλλον και να μην διακυβευτούν αυτές. Πώς εσείς θα συνεισφέρετε για την εδαφική συνοχή και ε, για τη στήριξη της εδαφικής συνοχής στην Ευρώπη μέσω των επενδύσεων. Υπάρχει μία μελέτη του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, ε, σύμφωνα με την οποία το ΕΦΣΙ θα μπορέσει να έχει την πλήρη, ε, την πλήρη ισχύ του σε χώρες όπου θα έχουν επίσης ε, εφαρμοστεί και συνοδευτικά μέτρα από το κράτος. Εσείς λοιπόν πώς θα συνεισφέρετε στην επιλογή συγκεκριμένων έργων τα οποία θα είναι ανεκτά και περιβαλλοντικά και κοινωνικά. Ο κύριος Εμπάσεϊκα, Ευχαριστώ κύριε και ευχαριστούμε για την εισαγωγική σας παρουσίαση. Για το Κοινοβούλιο, το ΕΦΣΥ είναι από τις σημαντικές προτεραιότητες για τη βελτίωση των επενδύσεων. Το γνωρίζετε. Ταυτόχρονα γνωρίζετε ότι το Κοινοβούλιο επέκρινε ενίοτε τη διαφάνεια και τη λογοδοσία της ε, ΕΤΕ. Και από αυτή την έννοια λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για μας και για τα δύο ζητήματα, τόσο η διαφάνεια σου και για τη λογοδοσία, να έχει καλύτερες επιδόσεις το ΕΦΣΥ από ότι η ΕΤΕ. Και θα σας ε, δώσω δύο συγκεκριμένα παραδείγματα που επικρίναμε την, το έργο Κάστορ αποθήκευση φυσικού αερίου στην Ισπανία και το Πασάντα Τιμέστρου, ε, υποδομή στην Ιταλία, έργο υποδομή στην Ιταλία. Εκεί πέκρινε το Κοινοβούλιο τα ζητήματα αυτά, υπέβαλε έκθεση στην ΕΤΕ, η οποία ουδέποτε απάντησε. Οπότε το ερώτημα μου προς εσάς είναι το εξής. Πώς θα έχει καλύτερες επιδόσεις το ΕΦΣΥ όταν θα χρειάζεται να απαντήσει τέτοια ερωτήματα του Κοινοβουλίου. Ή μάλλον θεωρείτε ότι μπορεί να χρηματοδοτούνται τέτοια έργα μέσω του ΕΦΣΥ. Ποιε θα είναι οι διαφορέ δηλαδή μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του ΕΦΣΥ. Ευχαριστώ κύριε Μάρτερα. Πρώτα απ' όλα, ο κανονισμός αυτός απαντά και την ερώτησή σας ε, για τους τομείς και η κοινωνική υποδομή σίγουρα είναι επιλέξιμος τομέας. Η κοινωνική στέγαση, για παράδειγμα, η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η απόκτηση δεξιοτήτων είναι πολύ σημαντική τομείς, οπότε και η κοινωνική υποδομή θα είναι κομμάτι αυτού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Ποια θα είναι όμως τα κριτήρια δεν μπορώ παρά να επαναλάβω αυτά που είπα. Κοιτάξτε τι επιτύχατε με τι διαπραγματεύσει ω κοινοβούλιο για τον πίνακα αποτελεσμάτων, για το scoreboard, διότι το scoreboard δεν είναι απλά... Ε, δεν αφορά απλά την κλασική τεχνική βιωσιμότητα ενό έργου, αφορά και του στόχου πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. αφορά και τι κοινωνικέ ε, επιπτώσει των έργων. Ο πίνακα αυτό βαθμολογία αποτελεί καθοδήγηση για την Επιτροπή Επενδυτικής πολιτική και καλύπτει επίσης οικονομικά, τεχνικά ζητήματα αλλά και ζητήματα όπως αυτά που μόλις αναφέρατε. Αυτός λοιπόν ο πίνακας αποτελεσμάτων θεωρώ ότι είναι μεγάλη πρόκληση, κάτι δύσκολο να γίνει, αλλά βασικός προσανατολισμός. Τώρα όσον αφορά την πτυχή της συνοχής, όπως ανέφερα προηγουμένως, θα πρέπει να υποστηρίζουμε τα έργα διαφορετικά ανάλογα με την περιφέρεια ή τη χώρα και να υποχρεωμαστε να αποφύγουμε οποιαδήποτε συγκέντρωση σε συγκεκριμένες χώρες ή τομείς. Αλλά μην φαντάζεστε ότι υπάρχει μία ενιαία λύση για όλους. Η Ρουμανία έχει άλλες ανάγκες από τη Φιλανδία, για παράδειγμα. Οι τομεί διαφέρουν. Σε ορισμένε χώρε έχουμε προηγμένε κεφαλαίε αγορέ και αλλού δεν υπάρχουν καν κεφαλαίε αγορέ. Εκεί θα λειτουργήσει καταλητικά το ΕΦΣΥ. Αλλού υπάρχουν ε, τράπεζες πρότσης, αλλού τώρα οικοδομούνται. Οπότε αυτή η ευελιξία είναι απόλυτα ε, σημαντική. Όσον αφορά τη διαφάνεια, επίσης εκεί ο κανονισμός αναφέρει σαφώς ότι υπάρχει ένα σύστημα υποβολής εκθέσεων αφενός, αλλά απ' την άλλη τα θεσμικά όργανα πρέπει να απαντούν, να δίνουν συγκεκριμένες απαντήσεις και αυτό θα το ελέγχει ο Γενικός Διευθυντής θα πρέπει να υποχρεώται να απαντά τι ερωτήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για μένα αυτό είναι απολύτως σαφέ. Υποχρεούμε να το πράξω. Δεν είναι απλά υποχρέωση. Είναι ο φυσιολογικός τρόπος συνεργασίας με έναν σημαντικό ε, ευρωπαϊκό εταίρο, ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο, ε, τόσο σημαντικό όσο το Κοινοβούλιο. Δεν έχω να δώσω απάντηση για το κατά, κατά πόσο υπάρχει απάντηση για τα θέματα Κάστρο και, του Μέστρε από την ΕΤΕΚ. Γνωρίζω τα έργα και τα θέματα που προέκυψαν για αυτά. Αν υπάρχουν αιτήματα για έργα του ΕΦΣ από το Κοινοβούλιο, ο Γενικός Διευθυντή υποχρεούται να απαντήσει. Ευχαριστούμε για το EFDD ο Μαρκοτζάνη. Ναι, ευχαριστώ. Ήθελα να ξαναπάμε στην πτυχή της προσθετικότητας που είναι πολύ σημαντική. Όπως αναγραφτέ σαφώς ε, στον κανονισμό θα είναι σημαντικό καθήκον τόσο του Γενικού Διευθυντή όσο και της Επιτροπής ε, Επενδύσεων. Εγώ είδα ότι τους τελευταίους μήνες, τις τελευταίες εβδομάδες η ΕΤΕ άτυπα έχει εγκρίνει έργα τα οποία ενδεχομένω θα χρηματοδοτηθούν ε, μέσω εγγύησεων του ΕΦΣΥ. Όσον αφορά αυτά τα έργα, τα οποία θα γνωρίζετε, δεν έχουν αυτό το χαρακτήρα της προσθετικότητας. Πρόκειται για έργα εταιρικής σχέσης με περιφερειακές ή τοπικές τράπεζες. Σκέφτομαι τώρα τη συμφωνία με το Κρέτο Εμιλιανό στην Ιταλία, με το μικροκρέτο Τρέντινο στην Ιταλία ή με την Bank στην ε, Γερμανία και έχω την εντύπωση ότι πρόκειται για συνήθεις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται χαλάρα μέσω προγραμμάτων που ήδη υπάρχουν ε, ε, μέσω της ΕΤΕ. Ήθελα να πείτε εσείς προσωπικά πώς ε, αξιολογείτε τα έργα αυτά. Πώς εσείς ως Γενικός Διευθυντής θα διασφαλίσετε ότι θα πληρείτε αυτό το κριτήριο της προσθετικότητας, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Και από αυτά τα πρώτα έργα που έχει ανακοινώσει η ΕΤΕ δεν φαίνεται να ε, υπάρχει αυτό το χαρακτηριστικό. Κύριε Βάλλη ναι, και εγώ θέλω να αναφερθώ στη διαφάνεια. Είναι θεμελιώδη στοιχείο. Διότι αυτό το ταμείο θα χρηματοδοτεί μεγάλα έργα και διακρίνουμε ένα πρόβλημα διαφάνειας και ενημέρωσης όσον αφορά τους διαγωνισμούς. Θέλουμε να μας πείτε κατά πόσο εσείς είστε διατεθειμένος να συνεργαστείτε στο μέγιστο, γιατί σε πολλές περιπτώσεις εμείς έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν δυσκολίες να λάβουμε τέτοιες πληροφορίες. Ενδεχομένως άμα τις θέλετε και εκ των προτέρων να μπορούν να αποφευχθούν ε, αμφιβολίες και αμφισβητήσεις. Θέλουμε λοιπόν μια εγγύηση απόλυτης διαφάνειας των πληροφοριών που αφορούν τα έργα. Ευχαριστώ. Κύριε Μόλτερε. Να πω ότι συμφωνώ απόλυτα ως προς το ότι η προσθετικότητα είναι στον πυρήνα εγχειρήματο, όπως προείπα. Πρέπει να προσθέτει κάτι στα εφιστάμενα προϊόντα με προφίλ ψηλού κινδύνου και όλα αυτά που προανέφερα. Είναι όλα σημαντικά αυτά, πράγματι. Δεύτερον, να διευκρινίσω ότι ναι, διατέλεσα αντιπρόεδρος της ΕΤΕΠ. Μέχρι τα τέλη Αυγούστου ήμουν αντιπρόεδρος. Πρώτα παραιτήθηκα όπως όφυλα αλλά πολύ νωρίτερα δεν συμμετείχα στις ε, διαδικασίες λήψεως ε, αποφάσεων ε, από τη στιγμή δηλαδή που έθεσε αποψηφιότητα έπρεπε να παραμείνω εκτός. Αρχικά το όλο εγχείρημα είναι έχει ως στόχο το συμφέρον και το όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Και αν δείτε και τη χρονική στιγμή το timing, 22 Ιουλίου αποφασίστηκε, αν θυμάμαι καλά, το ΕΦΣΥ. Εσεί, στο Κοινοβούλιο αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητήσατε από την ΕΤΕΠ πολύ απλά να ξεκινήσει ε, την όλη διαδικασία ακόμη και πριν συγκροτηθεί επίσημα ε, η Επιτροπή Επενδύσεων. Άρα έχουμε έργα τη ΕΤΕΠ και αποφασίζει την επικύρωση τη εγγύηση η Αυτή είναι η κατάσταση. Συμφωνώ ότι εμείς στο ΕΦΣΥ θα πρέπει να αναπτύξουμε περαιτέρω αυτά τα προϊόντα. Μίλησα για το equity, τα ιδιωτικά κεφάλαια που είναι ένα νέο πρόγραμμα, σημαντικό. Διαμοιρασμό κινδύνων, risk sharing, ε, μικροχρηματοδότηση, ε, και αυτό σημαντικό. Άρα ναι, εδώ είναι αφετηρία αυτή της διαδικασίας του warehousing, δεν είναι όμως και ο τερματισμός. Βρισκόμαστε απλά στην αρχή και με τις Εθνικές Αναπτυξιακές τράπεζε και του φορείς θα συνεργαστούμε και όλα αυτά ανοίγουν νέου οριζοντές. Ξεκινήσαμε στο πλαίσιο της ΕΤΕΠ με βάση το αίτημα και του Κοινοβουλίου την όλη διαδικασία. Δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε την προσέγγιση business as usual, να είστε βέβαιοι γι' αυτό, σε ό,τι τώρα τη διαφάνεια. Εγώ πρέπει να τηρώ τον κανονισμό τελεία και παύλα. Τον κανονισμό τον έχετε αποφασίσει εσείς νομικά εσεί είστε και εγώ δεσμεύονται από τι νομικές απαιτήσει. Αυτό είναι το μόνο το οποίο μετράει. Και ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να απαντά τι ερωτήσεις ε, όπως τις έχει δει μπροστά του, γραμμένες. Ε, εγώ είμαι πεπισμένο όμως και ουσιαστικά ότι η συνεργασία μαζί σας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για να στεφθεί με επιτυχία το εγχείρημα. E το ΕΝΕΦ e δεν βλέπω κανέναν συνάδελφο, λέει ο Πρόεδρος. Σας δώσω λοιπόν τώρα το λόγο για τις ε, καταληκτικές σας παρατηρήσεις. Να σας ευχαριστήσω καταρχάς ε, για την πολύ ανοιχτή και επικοδομητική αυτή συζήτηση. Γνωρίζω που υπάρχουν ε, ίσως προβλήματα, τι ενδιαφέρει το κοινοβούλιο, το έχω δει και στη των διαπραγματεύσεων και γνωρίζω ότι ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για συγκεκριμένα. Όλα αυτά τα αντιλαμβάνουμε και τα γνωρίζω πλήρως. Αυτό το οποίο είπα είναι ότι εμείς στο Ταμείο Στατικών Επενδύσεων ε, στη διοίκηση κάνουμε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στεφθεί με επιτυχία αυτό το εγχείρημα. Και αυτό μπορεί να γίνει με τη δική σας υποστήριξη. Και αυτή η επικοινωνία είναι πάντα αμφίδρομη, ποτέ μονόδρομος και γι' αυτό ε, θα παλέψω και έχω εμπιστοσύνη και στην ότι θα έχω την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να στεφτεί με επιτυχία προς όφελος των Ευρωπαϊκών πολιτών το ΕΦΣΥ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ακρόαση, για τις απαντήσεις σας και μπορούμε τώρα να περάσουμε στην κυρία Τσάνοβα και δίνω το λόγο στον Ζαν. Ευχαριστώ Ρομπέρτο να καλέσω την κυρία Ηλιάνα Τσάνοβα να έρθει εδώ στην έδρα. Το όνομά σα, αξιότιμη κυρία, μας το κοινοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο ε, για την ασκή τη αναπληρώτρια γενική Διευθύντρια. Έχετε πέντε λεπτά για μια εισαγωγή. Παρακαλώ, καθίστε. Και έχετε το λόγο. Thank you very much, Mr. Chairman. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής, ε, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε εδώ για να σας μιλήσω. Είναι δύσκολο για μένα να σταθώ στο ύψος του κυρίου Μάλτερερ και να μην επαναλάβω τα εκπληκτικά πράγματα που είπε κατά την παρουσίασή του. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω την ιδιαίτερη εκτίμησή μου για το δικό σας έργο μέχρι σήμερα όσον αφορά το ΕΦΣΙ. Παρακολουθώ στενά τη διαδικασία και πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί από το τεράστιο έργο που έχει επιτευχθεί από τη Συμβουλή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Έχω μεγάλο σεβασμό για σας. Για μένα είναι τιμή και προνόμιο που βρίσκομαι εδώ απόψε ως υποψήφια για αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του ΕΦΣΥ. Και θα σας παρουσιάσω το επαγγελματικό μου υπόβαθρο, εν συντομία, η σταδιοδρομία μου σε μεγάλο βαθμό αφιερώθηκε στις αναπτυξιακές τραπεζικές συναλλαγές. Πάνω από 12 χρόνια τα πέρασα σε έναν οργανισμό παρόμοιο, οργανισμό με την ΕΤΕ, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα ε, ε Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης, ε, ε, υπεύθυνοι για έργα που περιλαμβάνονται και στην καρδιά του κανονισμού ΕΦΣΙ σε νεότερα κράτη-μέλη που είναι λιγότερα αναπτυγμένα σε σχέση με τα άλλα. Επίσης, ε, χρηματοδότησα έργα ε, με υψηλότερο βαθμό κινδύνου, κάτι που επίσης χαρακτηρίζει το ΕΦΣΙ, οπότε θεωρώ ότι η εμπειρία μου θα συμπληρώσει επικοδομητικά ε, τις υπάρχουσες δυνατότητε της ΕΤΕ ώστε να είναι επιτυχή τα έργα αυτά στο μέλλον. Όπως βλέπετε από το βιογραφικό μου είχα και την τιμή να βοηθήσω τη χώρα μου δύο φορές σε περίπτωσης κρίσης ως ε, υφυπουργό για τη διαχείριση ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. Ε, στην μεταβατική κυβέρνηση είχα απέκτησε εμπειρία όπου είδα προκλήσεις ε, για τις οικονομίες των χωρών αυτών που έχουν πληγεί από κρίσεις ε, οικονομική αστάθεια, ε, ρυθμιστική αβεβαιότητα και λοιπές περιπτώσεις αβεβαιότητας. Και γνωρίζω από τη δική μου εμπειρία ότι ένα μέσο όπως το ΕΦΣΥ πραγματικά θα μπορούσε να σημαίνει μια διαφορά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μόνο εάν υλοποιηθεί σωστά. Τι εννοώ. Πρώτα απ' όλα, η εγγύηση του ΕΦΣΥ πράγματι θα υποστηρίξει έργα που χρειάζονται τις απαιτήσει προσθετικότητας του κανονισμού και θα υποστηρίξει έργα που θα αποδείξουν την πρόσθετη αξία όσον αφορά την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην επιτρέψουμε υπερβολικά τομεακή ή εδαφική συγκέντρωση έργων. Και όπως είδα αυτό είναι θέμα που ανησυχεί και εσάς. Εδώ να προσθέσω ότι θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να υπάρχει σωστή προετοιμασία των έργων όχι μόνο στα κράτη-μέλη που έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τέτοια έργα αλλά και στα κράτη-μέλη τα οποία χρειάζονται επιπλέον στήριξη για να προετοιμάσουν έργα καλής ποιότητας. Όπως είπε και ο κύριος Μορτερέρ, το ΕΦΣΙ ανήκει σε ένα ευρύτερο σχέδιο για την Ευρώπη και η επιτυχία του θα εξερθεί σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική ηγεσία και τη βούληση των κρατών μελών και της Επιτροπής για υλοποίηση των κρίσιμων μεταρρυθμίσεων ώστε να άρουμε τα εμπόδια ε, προς τι ιδιωτικέ επενδύσει και την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε φάση όπου πρέπει να θέσουμε σε λειτουργία το ΕΦΣΙ ώστε να εκπληρώσουμε του στόχου που αναφέραμε. Και ξεκινάμε από την Επιτροπή Επενδύσεων και τα μέλη τη. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται ότι μέσα στου επόμενου δύο μήνε τα οκτώ μέλη τη Επιτροπή Επενδύσεων θα έχουν διοριστεί. Μια σειρά λειτουργικών κατευθυντηρίων γραμμών και διαδικασιών ακόμη βρίσκονται υπό μελέτη και θα καθορίσουν το ρόλο ε, της διακυβέρνησης του ΕΦΣΥ σε σχέση με τα τμήματα των εταίρων της με τα οποία θα συνεργάζεται. Επίσης ε, έχω πει και με τον κύριο Μολτέρο ότι πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο τον ιδιωτικό τομέα για τις δυνατότητες που προσφέρει το ΕΦΣΥ ώστε όχι μόνο να κινητοποιήσουμε ιδιωτικά κεφάλαια αλλά και να αυξήσουμε τον αριθμό συμμετεχουσών ιδιωτικών εταιριών. Uh, Εάν λάβω τη θέση της αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας θα προσπαθήσω να διευκολύνω ανοιχτό και διαφανή διάλογο μεταξύ των κύριων ενδιαφερομένων όπως της ΕΤΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίως και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μια άλλη πτυχή της εργασίας μου θα είναι συντονισμός ε, στο εσωτερικό και της ΕΤΕ και θα σταματήσω εδώ και θα ήθελα να ακούσω τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία μου. Θα έχετε τη δυνατότητα και στη δευτερολογία σας αλλά και απαντώντας ε, στα ερωτήματά μας να δώσετε απαντήσεις. Πρώτος ο κύριος Φερνάντης για να κάνει ερώτηση για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω και εγώ την υποψήφια και να πω πως εντυπωσιάστηκα από τα επιτεύγματα της μέχρι τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως και εσείς ελπίζω, ενδιαφέρεται πάρα πολύ να υπάρχει συνέργεια ανάμεσα στο ΕΦΣΙ και στα άλλα ε, μέσα. Μπορεί να επιτευχθεί συνεργασία μέσω μιας επενδυτικής πλατφόρμας ε, ή κάπως έτσι. Εσείς ε, πώς ε, σκοπεύετε να στηρίξετε αυτές τις ε, συνέργειες και να προωθήσετε λοιπόν αυτήν την πολυπόθητη ισορροπία στις επενδύσεις. Πώς μπορείτε να αντλήσετε από τη δική σας εμπειρία έτσι ώστε να συνεισφέρετε στην επίτευξη των συνεργειών ανάμεσα στις, ε, στις επενδύσεις, ιδιωτικούς επενδυτές και το ΕΦΣΥ. Έχετε δύο λεπτά για να απαντήσετε δύο δυόμιση λεπτά, όχι γιατί ο εισηγητή πρέπει να λάβει άμεσα απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματι πιστεύω πως ε, υπάρχει μεγάλο περιθώριο άλληλος πλήρωσης ανάμεσα στο ΕΦΣΙ και στις επενδύσεις, ιδιαίτερα σε χώρες που έχουν τεράστια επενδυτικά κενά και το ΕΦΣΙ δεν αρκεί για να καλύψει τις επενδυτικές τους ανάγκες. Εκεί λοιπόν βλέπω πως υπάρχει μεγάλο δυναμικό για, προ... για συμπληρωματικότητα, όχι μόνο για μεγάλα έργα υποδομών, αλλά και για μικρότερα έργα που θα στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μικροδανισμός, για παράδειγμα, δημιουργία πλατφόρμανς που θα αναλαμβάνει τον κίνδυνο και θα δώσει έτσι την δυνατότητα σε άλλους επενδυτές όπως την ΕΤΕ, τον ιδιωτικό τομέα, τις εθνικές ε, τράπεζες να ε, συνεισφέρουν. Θα συγκεντρώσουμε λοιπόν χρηματοδότηση από διάφορες πηγές και το ΕΦΣΙ σκοπεύει να αναλάβει τη, τους μεγαλύτερους κινδύνους στην χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ούντο Μπούλμαν. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε κυρία Τζάνοβα. Εργαστήκατε για την Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης που είναι έτσι ένας ανταγωνιστικός θεσμός ε, προς την ΕΤΕΠ. Κάτι που δεν είναι φυσικά κατά ανάγκη εμπόδιο μπορεί αντιθέτως να μας ε, δώσει νέα επιχειρήματα και να δώσει όθηση σε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Αν δούμε τις υφιστάμενες πρακτικές της ΕΤΕ, πώς επιλέγει δηλαδή έργα, πώς τα αξιολογεί και εάν το συγκρίνουμε αυτό με τις ε, νέες υποχρεώσεις που δημιουργεί ο κανονισμός ΕΕΣΥ, εσείς ποια νομίζετε πως είναι η κυριότερη διαφορά, τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά ως προς την επιλογή των έργων για χρηματοδότηση σύμφωνα με τον κανονισμό, πώς εσείς ερμηνεύετε τον πίνακα επιδόσεων πάλι σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕΣΥ, και σχετικά με αυτό το μείγμα πολιτικής, έργων και γεωγραφικής κατανομής αυτών. Ε, να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει και το παράρτημα 2 του κανονισμού, το οποίο δίνει τη δυνατότητα ε, στο Διοικητικό Συμβούλιο να αναλάβει την επιλογή των έργων και να δημιουργήσει σε γραμμές για την γεωγραφική και τομεακή κατανομή. Εσείς, τι θα συστήνατε στο Διοικητικό Συμβούλιο, θα του συστήνατε να χρησιμοποιήσει αυτή την ευκαιρία για να λάβει νέες ε, επιλογές, για νέους ε, τομείς κατανομής των έργων αυτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα έχετε απόλυτα δίκιο. Η ΕΤΕ θα χρειαστεί να αναπροσαρμόσει την οτροπία της ώστε να μπορέσει να υλοποιήσει το εύση επενδύοντας σε έργα υψηλότερου κινδύνου σε σύγκριση με τον συνήθι κινδύνο που λαμβάνουν από τις δικές μου συζητήσεις μαζί τους το γνωρίζουν απόλυτα και υιοθετούν μέτρα ώστε να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του κανονισμού. Εγώ θα συνεργαστώ στενά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παρέχοντας και τη δική μου εμπειρία και βάσει του σημερινού θεσμικού πλαισίου που έχουμε ώστε να ευνοήσουμε έργα υψηλότερου κινδύνου. Όσον αφορά τον πίνακα αποτελεσμάτων και τις απαιτήσει, το περιβάλλον στο οποίο ζούμε είναι ταχαίως εξελισσόμενο. Δεν αποκλείω αφού αρχίσει να λειτουργεί το έύση και δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα, δεν αποκλείω να προσαρμόσουμε κάποιες από αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές ώστε να ταιριάζουν καλύτερα με τις σημερινές συνθήκες της αγοράς. Εγώ όταν ε, ήρθα σε επαφή με το Διοικητικό Συμβούλιο και με την ΕΤΕ συμφωνήσαμε ότι θα χρειαστεί να δείξουμε ευελιξία και να προσαρμοζόμαστε στις ε, συνθήκες της αγοράς. Τρία χρόνια είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στους κοιόδης εισηγητές. Δύο ανά ομάδα, μισή λεπτό, ο κάθε σκιώδης. Ο Κάρας, καταρχάς. Θα είμαι απολύτως ειλικρινής. Χαίρομαι πάρα πολύ για το ότι δεν προαρχίστε ούτε από την ΕΤΕ, ούτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά φέρνετε ένα νέο άνεμο και νέες εμπειρίες ε, μαζί σας. Έχετε λοιπόν εμπειρία εργαζόμενη στη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και ε, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ήσασταν αρμόδια για την δημιουργία και ανάπτυξη υποδομών. Ε, και ήσασταν στο Λονδίνο πιο πριν στην πρώην Ιουκοσλαβία, στην ε, Βουλγαρία και μετά ήρθατε εδώ. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιες είναι οι εμπειρίες που αποκομίσατε από όλα αυτά τα μέρη που εργαστήκατε, που θα μπορέσετε να τη χρησιμοποιήσετε στην, ε, στο επιχειρησιακό σχέδιο της, ε, του ΕΦΣΥ. Δεν αναγράφονται ακριβώς οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή στο καταστατικό του ΕΦΣΙ και ποια είναι η διαφορά λοιπόν μεταξύ της δικής σας ε, θέσης ε, και της θέσης του Γενικού Διευθυντή και ποιες είναι οι προτεραιότητες που έχετε θέσει για ε, εσάς και για το έργο σας εκεί. Ο κύριος Μούρεσεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η πρώτη μου ερώτηση σχετίζεται με την τελευταία ερώτηση του συναδελφού Ατμαρκάρας για το δικό σας ρόλο και τις ευθύνες σας και η ερώτησή μου είναι η Προβλέπετε ότι θα έχετε δικό σας χαρτοφυλάκι ευθυνών από την πρώτη μέρα ή αναμένετε να σας εκχωρούνται προνόμια και ευθύνες από το Γενικό Διευθυντή. Και η δεύτερη μου ερώτηση είναι ποια στρατηγική, ποιες προτεραιότητες έχετε στο νου σας για τη διάδοση των πληροφοριών σε σχέση με το ΕΦΣΥ. Θα προσπαθήσετε να προσελκύσετε ε, ακολούθως ε, περαιτέρω ε, πιθανούς επενδυτές στο ΕΦΣΙ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα για να απαντήσω στον κύριο Κάρας. Από τη δική μου εμπειρία ως ε, τραπεζίτη ε, πιστεύω έμαθα πράγματα που σχετίζονται με το στεγενούς στο ΕΦΣΙ. Χρηματοδοτούσαμε έργα πολύ υψηλή προστιθέμενης αξία για την οικονομική ανάπτυξη των εν λόγω χωρών. Οπεργάστηκα, εργάστηκα στρατηγικέ στρατηγικές υποδομές, αστική ανάπτυξη, ενεργειακή απόδοση. Πολύ συχνά χρειάστηκε να προωθήσω περισσότερε καινοτόμε ε, λύσει, κάτι που μοιάζει με τη δομή του ΕΦΣΥ κινητοποιώντας ε, δημόσιου πόρους ε, βαστών οποίων προσελκύα με ιδιωτικές επενδύσεις από εταιρείε ή τράπεζε, στοχεύοντα ε, τομεί που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα στην αγορά. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι έχω τις ικανότητες ε, στη νέα μου θέση να χρησιμοποιήσω την εμπειρία που απέκτησα τα τελευταία χρόνια και να συμβάλλω στην επιτυχία του ΕΦΣΙ. Επίσης, ε, όπως είπα, έχω χρηματοδοτήσει έργα πολύ υψηλότερου σε επικινδυνότητας από ότι χρηματοδοτεί μέχρι στιγμής ε, η ΕΤΕ. Οπότε με μεγάλη μου χαρά να μοιραστώ την εμπειρία μου με την Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ τώρα που πρέπει να προσαρμόσουμε τους κανόνες διαχείρισης κινδύνου για το ΕΦΣΥ. Πώς βλέπω εγώ τα δικά μου καθήκοντα. Συνάντησα τον κύριο Μόλτερ μόλι χθε. Οπότε δεν έχουμε ακόμα καθίσει να συζητήσουμε πώ θα οργανωθούμε. Ε, Κάποιο είπε ότι ο Γενικό Διευθυντή είναι ο υπουργό Εξωτερικών και ότι ο αναπληρητής ε, ε, Γενικός είναι ο υπουργό Εσωτερικών. Οπότε θα προσπαθήσω να διευκολύνω τον εσωτερικό συντονισμό μεταξύ των επιχειρησιακών ομάδων τη, ΕΤΕ, αφενό οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του ΕΦΣΥ και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΣΙ, από την άλλη που θα έχουμε το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επενδυτική Επιτροπή. Οπότε αυτέ θα είναι η πρώτη μου προτεραιότητα. Να υπάρχει ομαλή λειτουργία και συνεργασία μεταξύ αυτών των δύο οργάνων. Δεύτερη προτεραιότητα, να ξεκινήσουμε το ταχύτερο δυνατόν με τις Εθνικές Τράπεζες Πρόθεσης γιατί πρέπει να βρούμε έναν τρόπο συνεργασίας ώστε να δραστηριοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν. Αυτό πιστεύω δεν απάντηση και στη δεύτερη ερώτηση διότι πρόκειται για σημαντικά πράγματα και θα μάθουμε τα υπόλοιπα στην πορεία. Ευχαριστώ. Um, σας ευχαριστώ πολύ εκ μέρου ε, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η Αίντερ Γκαρτία Θάπελ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε και την κυρία Τσάνοβα στην Επιτροπή Προπολογισμών αλλά και στο Κοινοβούλιο Εν Γέννη. Ένας από τους ε, μεγαλύτερους φόβους ε, και κριτικές που ασκούσαμε σε αυτό το ταμείο ήταν ότι είχαμε τα 8 δις που τα παίρνουμε από τον προπολογισμό και τα βάζουμε στην Τράπεζα Επενδύσεων όπως είδαμε και ένα από τα πρώτα μας κριτήρια είναι πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα θα μιλάμε για μια απλή μεταφορά πιστώσεων, αλλά θα χρηματοδοτηθούν και θα γίνουν άλλα έργα που δεν θα γίνονταν αν δεν υπήρχε το ΕΦΣΥ. Πώς αυτό θα εξασφαλιστεί αυτή η προσθετικότητα δηλαδή. Και επίσης αυτά τα κριτήρια οικονομικής συνοχής και κοινωνικής συνοχής, πώς θα ε, είναι προτεραιότητα αυτά τα κριτήρια για την απόφαση περί χρηματοδότησης συγκεκριμένων έργων. Αυτό έχει να κάνει και με τη γεωγραφική κατανομή αλλά και με μια τομεακή αν θέλετε κατανομή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, έχει ε, ορίσει κάποιους τομείς ως τομείς προτεραιότητας για την χρηματοδότηση. Πώς πιστεύετε εσείς ότι θα κριθεί η επιτυχία αυτού του ταμείου με την τομεακή εφαρμογή, για παράδειγμα, ενεργειακή απόδοση είναι ένα από τα πάγια αιτήματα του Κοινοβουλίου. Εσείς πώς πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει επιτυχία με έργα ενεργειακή απόδοση, εφόσον είπατε ήδη ότι έχετε εργαστεί κατά το παρελθόν σε αυτό το τομέα. Τι μπορεί να προσφέρει σε αυτό το τομέα ή σε οποιονδήποτε άλλο το Ταμείο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο Μιγελίζα φεραιρα Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο μου ερώτημα να έχουμε έτσι μια πιο αναλυτική προσέγγιση για τα έργα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια έργα που είναι στην λεγόμενη αποθήκη της ΕΤΕΠ και ενέχει ε, κάποιο κίνδυνο ε, το έργο όταν έχουμε συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων, εκτός ένωσης δηλαδή. Εσείς πώς θα αντιμετωπίζατε αυτό ή άλλα παρόμοια ζητήματα αν δεν υπάρχει πλήρη συμμόρφωση με τους κανονισμούς, ε, θα στραφείτε εναντίον ε, ή θα έχετε μια ευρεία ερμηνεία της εντολής σα. Δεύτερον, από την εμπειρία σας, που είναι καλή εμπειρία σας, έχετε εργαστεί όμω κυρίω ε, σε ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες και νέοι ερχόμενες στην Ένωση τι θα λέγατε για την οικονομική κατάσταση στην Ευρωζώνη και σε άλλες περιοχές όπου εξακολουθεί να μαστίζονται από τεράστια κρίση, μεγάλο ε, αποπληθωρισμό. Και δεν είναι το ίδιο ε, αποφυγή σύγκλησης. Δεν θέλουμε και υπερβολική συγκέντρωση όμως από την άλλη πλευρά. Τέλος, αν έχω χρόνο για να κάνω μια τρίτη ερώτηση, η διαφορά μεταξύ των έργων αυτών σε σχέση με την προηγούμενη εμπειρία, BERD και αυτά που γνωρίζετε από την ΕΤΕΠ, τι διαφορές υπάρχουν σε αυτό το καινούριο έργο. First um, ε, για το στοιχείο της προστατικότητας να πω πως η προσέγγιση μας είναι δυτή, από όσο ξέρω μέχρι τώρα από τη μία να συνεργαζόμαστε πολύ στενότερα με τις Εθνικές Τραπεζές Προώθησης και από την άλλη και ο πίνακας επιδόσεων που έχει προστιθέμενη αξία, μας δίνει σαφείς ενδείξεις για την προστιθέμενη αξία του κάθε έργου. Όταν λοιπόν αξιολογούμε κάποιο έργο, θα είμαστε προσανατολισμένοι στον, είμαστε μάλλον μέχρι τώρα προσανατολισμένοι στον πίνακα επιδόσεων και στην αξιολόγηση. Εμείς πιστεύω στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΣΥ θα συνεργαστούμε σε πολύ ε, προηγούμενο στάδιο έτσι ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε καλύτερα τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν κάτω από το ΕΦΣΥ. Πώς θα κάνουμε το Ταμείο Επιτυχές. Πιστεύω πως είναι σημαντικό να αναπτύξουμε δράση το συντομότερο. Ξέρω πως πολλές χώρες έχουν προτείνει ίδιες κάποια έργα όμως γνωρίζω επίσης πως και αυτά τα έργα, αρκετά από αυτά έστω, δεν είναι κατάλληλα για χρηματοδότηση από το ΕΦΣΙ. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει μια οργανωμένη προσπάθεια έτσι ώστε να επιλεγούν έργα τα οποία θα έχουν μεγάλη προστιθέμενη αξία στην ευρωπαϊκή οικονομία. Τώρα, με ρωτήσατε για τα ξένα κεφάλαια που θα επενδύσουν σε διάφορα έργα. Πιστεύω πως ε, πρέπει να το εξετάσουμε αυτό κατά περίπτωση. Δεν μπορούμε να έχουμε μία προσέγγιση για τα πάντα. Θα σας δώσω λοιπόν περισσότερες πληροφορίες όταν έχω στα χέρια μου συγκεκριμένα παραδείγματα τέτοιων έτσι, αμφιλεγόμενων έργων. Μία ερώτηση από την κυρία Φερέρια. Δηλαδή τι να περιμένουμε, να μην τα δεχτείτε ή ότι θα τα δεχτείτε. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Δεν μπορώ να απαντήσω γιατί είναι πολύ γενικό το ερώτημά σας. Χωρίς να ξέρω δεν μπορώ να απαντήσω. Εγώ θα εφαρμόσω τις απαιτήσει του κανονισμού ΕΦΣΙ και την πρώτερη επαγγελματική μου εμπειρία. Και μην ξεχνάτε πως υπάρχουν και συγκεκριμένες επιτροπές μέσα στο ΕΦΣΙ που λαμβάνουν και εκείνες ε, αποφάσεις. Και θα αξιολογήσουν αν μπορούμε να κάνουμε αποδεκτό ένα έργο για χρηματοδότηση ΕΦΣΥ ή όχι. Έχω πλήρη επίγνωση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν ε, όλες ε, οι χώρες και οι πιο ανεπτυγμένες. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και εξαιτίας της ε, κρίσης και δεν μπορούμε να τη λύσουμε αυτή χωρίς να αλλάξουμε προσέγγιση. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ελλείψεις στη ρίζα τους. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το επενδυτικό κοινό στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Μας τέλειωσε ο χρόνος, λυπάμαι. Ζητώ συγγνώμη για τους ECR και Swinburne. I will keep my questions very short, so there will be a little more time and you... Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη έτσι ώστε να έχετε χρόνο να απαντήσετε στις ερωτήσεις που δεν προλάβατε. Σας ευχαριστώ πολύ για τα εισαγωγικά τα σας σχόλια. Ε, η δική μου ερώτηση έχει να κάνει με την προσπάθειά μου να αξιολογήσω την καταλληλότητά σας για αυτόν τον ε, ρόλο. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας ε, λοιπόν θα φροντίσετε να συνάδουν οι στόχοι του ΕΦΣΙ με τα έργα. Θα πρέπει λοιπόν να να έχετε αναπτύξει κάποιες ικανότητες οι οποίες θα σας βοηθήσουν να κάνετε αυτόν τον ρόλο. Εσείς πώς θα διασφαλίσετε ότι η Επιτροπή Επενδύσεων θα εκτελέσει τις αρμοδιότητές της, θα παίξει τον ρόλο της. Από την άλλη να πω ότι πιστεύω πως έχετε τις ικανότητες να διοικήσετε ένα τέτοιο πάνελ, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω εάν έχετε πρώτερη εμπειρία σε αυτό. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλα μέλη του ECR που θέλουν να λάβουν το λόγο. Όχι, όλα υπόθηκαν για το ECR. Παρακαλώ. Για την απάντηση. Λοιπόν, η απάντηση είναι ναι. Έχω εκτενή εμπειρία διαχείρισης ε, ομάδας εμπειρογνωμόνων ε, που εργάζονται για έργα. Τα έργα στα οποία εργαστήκα εγώ ε, τα διαχειριστήκαν περίπλοκες ομάδες αυτή τη στιγμή προεδρεύω ένα επενδυτικό ταμείο για τα Δυτικά Βαλκάνια το οποίο διαχειρίζεται ένας διαχειριστής ε, ταμείου και είμαι και μέλος του Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε γνωρίζω τι ε, τις διάφορες συνιστώσεις ε, και τη δική μου λειτουργία. Σε περίπτωση που χρειαστεί δηλαδή να κάνω κάτι στη θέση του Γενικού Διευθυντή είμαι πεπισμένοι ότι μπορώ να εκπληρώσω τα καθήκοντά μου όσον αφορά τα έργα όπως είπαμε η Επιτροπή Επενδύσεων θα λαμβάνει τις αποφάσεις. Αυτό μπορώ να κάνω εγώ είναι να είμαι ανεκτόμυαλη και να συζητώ μαζί τους καθαρά και με διαφάνεια για τις δικές μου εντυπώσεις για τα έργα αυτά και να ανοίγω μια συζήτηση εκ των προτέρων ώστε να βλέπουμε κατά πόσο οι απαιτήσει του πίνακα αποτελεσμάτων πληρούνται και κατά πόσο μπορούμε να συνεχίσουμε με το έργο. Αλλά στο τέλο, τέλο, η Επενδυτική Επιτροπή θα είναι αυτή που θα λαμβάνει τι αποφάσει και όχι η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια. Ευχαριστούμε. Για το φιλελεύθερους, ο κύριος Ντεπρέ. Δεν είμαι εγώ, ο συναδελφός μου είναι, κύριε Πρόεδρε. Το μοιραζόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ για την εισαγωγή. Έχω δύο ερωτήσεις. Το ΕΦΣΥ δημιουργήθηκε για να απευθυνθεί και σε ιδιωτικό κεφάλαιο και εσείς έχετε υπόβαθρο σε ε, ε τράπεζες που είναι δημόσιου χαρακτήρου. Με τι στρατηγική λοιπόν εσείς θα προσελκύσετε αυτό το ιδιωτικό κεφάλαιο στο ΕΦΣΙ. Δεύτερη ερώτηση ε, ε, θέτω την ίδια και στον κύριο Μόλτερερ. Έχετε κάποιο υπόβαθρο σε δημόσια χρηματοδότηση, αλλά το μεγάλο κομμάτι των χρημάτων του ΕΦΣΥ βρίσκεται εκεί για υψηλότερου κινδύνου επενδύσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου, καινοτομία. Κανένας από εσάς βάσει του βιογραφικού σας δεν έχει τέτοια εμπειρία. Πώς θα το διαχειριστείτε, πώς μπορείτε να διασφαλίσετε ότι τα επενδυτικά κομμάτια που διαχειρίζονται ε, τα Ευρωπαϊκά Επενδυτικά Ταμεία και όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα επενδυθούν στους τομείς αυτούς που θα δημιουργήσουν τη μεγαλύτερη ε, πρόσθετη αξία για την ευρωπαϊκή οικονομία. Γιατί μιλάμε συνέχεια για δημόσιες επενδύσεις αλλά σε τελική ανάλυση τελικά το ζήτημα είναι να επενδύσουμε σε μεγάλο βαθμό και την ιδιωτική επένδυση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το ιδιωτικό κεφάλαιο. Σίλβι Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, αξιότιμη κυρία, χαίρομαι που βρίσκετε σκέστε εδώ. Πιστεύω ότι ένα ταμείο που θα επενδύσει στο μέλλον θα τύχει καλύτερη διαχείριση εφόσον τηρούμε την αρχή τη ε, ισότητα μεταξύ φύλων. Αλλά πρέπει να υπάρχουν και απαραίτητε γνώσει. Εγώ θέλω να επικεντρωθώ το ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο είναι ένα από του τομεί ε, όπου είναι πολύ δύσκολο να γίνουν επενδύσει, παρότι αυτέ οι επενδύσει είναι επίγουσε δεδομένε ειδικότερα τη κατάσταση σε ορισμένε χώρε, όπου παρατηρούμε ότι πολλοί είναι δεν βρίσκουν δουλειές. Πώς θα αντιμετωπίσετε λοιπόν τις επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Αυτό το συγκεκριμένο ερώτημα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, απαντήστε. Έχετε το λόγο να απαντήσετε. Thank Σας ευχαριστώ. Καταρχάς, για το κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου. Ε, απόλυτα δίκιο έχετε και όπως είπα και στι εισαγωγικές μου παρατηρήσεις πρέπει να καταβάλουμε πλέον προσπάθεια για να μπορούν ε, να προωθούν τα έργα ε, και είπατε ότι ζητούνται επενδύσεις επιχειρηματικού κινδύνου, venture capital, στον τομέα της καινοτομίας ιδίως, ε, το ΕΑΦ το εμπιστεύομαι, γιατί τα τελευταία χρόνια το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, κόσμε και άλλες πρωτοβουλίες. Ελπίζω λοιπόν ότι με τις υποδομές και το έξτρα κεφάλαιο του ΕΦΣΙ θα μπορέσουμε να καλύψουμε το επενδυτικό κενό της ανάγκης επένδυσης με υψηλού κινδύνου. Από την άλλη πλευρά. Γιατί θα πρέπει να καταβάλει παραπάνω προσπάθειες για, να, για τις επενδύσεις υψηλού κινδύνου και την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Αυτό έχει ξεκινήσει, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον. Θα πάρει κάποιο χρόνο, αλλά νομίζω ότι τους δύο-τρεις επόμενους μήνες θα έχουμε ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει στη τράπεζα να αναλαμβάνει και τις επενδύσεις ε, ιδιωτικών κεφαλαίων. Ανάγκη επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Πολύ σωστό και πράγματι και η εκπαίδευση και η μικροχρηματοδότηση είναι από τους επιλέξιμους τομείς στο πλαίσιο του ΕΦΣΥ. Δεν είναι ξεκάθαρο βέβαια το κατά πόσο θα έχουμε σαφή ε, ζήτηση για τέτοιου είδους έργα. Και αν όχι, νομίζω ότι θα πρέπει να συγκεντρώσουμε και τις προσπάθειές μας. Να έχουμε δηλαδή μια δεξαμενή τέτοιων έργων ε, στο Συμβουλευτικό Κέντρο. Ευχαριστώ. Λέω πρόεδρος από την ομάδα Good. Ριάντα. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη κι εγώ. Πώς σχεδιάζετε να αντιμετωπίσετε ε, κράτη-μέλη που δεν έχουν ε, παρουσιάσει στο δημοστραπεζικό τομέα επαρκή πρόοδο ε, και για τις ΜΜΕ και τι ρόλο βλέπετε για τις ιδιωτικές τράπεζες ως SPVs. Κύριος Δεμάζη. Κύριε Τσάνοβα, είπατε νωρίτερα ότι θα εξετάζετε κάποια έργα κατά περίπτωση. Αν έμαθα σωστά, έχουμε το παράδειγμα των επιπτώσεων στα επιδετικά ταμεία ε, παγκόσμιας γεωγραφικής ε, εφαρμογής. Αλλά εδώ υπάρχουν κίνδυνοι να υπάρξουν απώλειες κάπου αλλού και να υπομειστούν το βάρος οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι. Οπότε πείτε μου, ε, κρίνοντας κατά περίπτωση, πώς θα αντιμετωπίζατε μια τέτοια απόφαση. I'm not aware of... Δεν γνωρίζω το συγκεκριμένο έργο που αναφέρατε, όμως πιστεύω πως είναι ζήτημα αρχής οι εγγυήσεις του ΕΦΣΙ να καλύπτουν μόνο κινδύνους οι οποίοι θα σχετίζονται με έργα εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι να καλύπτουν κινδύνους από έργα που προέρχονται από άλλες αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν δεν θεωρώ πως είναι σωστό να καλύπτονται κίνδυνοι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε περίπτωση κάποιας διασυνοριακής ε, συνεργασίας. Πιστεύω πως παρόλα αυτά, ακόμα και σε αυτά τα έργα, είναι σημαντικό να δούμε ποια είναι η προστιθέμενη αξία για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη, για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης κτλ. κτλ. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο να κρίνω κάτι χωρίς να ξέρω τις ε, συγκεκριμένες ε, λεπτομέρειες. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να επιτρέψω την εγγύηση του ΕΦΣΙ να καλύψει κινδύνους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός των 28 κρατών μελών. Εντάξει και φυσικά ε, αναφέρομαι και στην περίπτωση κάποιας συνοριακή ε, συνεργασία. συνεργασία. Τώρα ποιες δημόσιες τράπεζε, δηλαδή ε, έχετε υπόψη. Ναι, στην Ιρλανδία δεν έχουμε κάποιο δημόσιο τραπεζικό σύστημα στο οποίο μπορούν να καταφύγουν οι μικρομέσες επιχειρήσεις για να ζητήσουν χρηματοδότηση. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω εάν εσείς έχετε κάποια πρόταση έτσι ώστε να διασφαλίσετε την πρόσβαση αυτών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ε, χρηματοδότηση, όπως γίνεται στη Γερμανία για παράδειγμα. Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις ε, πιστεύω πως η λύση είναι απλή. Χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες ε, δομές, εγγύησεις για το μικροδανεισμό για παράδειγμα, μπορούμε να μοιραστούμε τον κίνδυνο ή να τους παρέχουμε ρευστότητα. Τώρα, μικροχρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εδώ να σας πω ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποιο, κάποια, κάποιο δημόσιο σύστημα χρηματοδότηση, τραπεζικό σύστημα. Μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από άλλες πηγές εκτός από τις τράπεζες. Γιατί φυσικά μια τράπεζα χρειάζεται να λειτουργεί και σωστά και καλά για να μπορέσει να παρέχει αυτή την βοήθεια, την ρευστότητα, χρηματοδότηση. Για τους πρασίνους, ο κ. Μαραγκάλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Τσάνοβα, ακούσαμε τον κύριο Μόρτερερ πριν από εσάς ε, που σε κάποιο βαθμό εκπροσωπεί τη συνέχεια, την κουλτούρα ΕΤΕΠ δηλαδή. Και τον κίνδυνο βέβαια που ενέχει αυτή η συνέχεια. Εσείς εκπροσωπείτε το νέο, το καινούριο. Αυτό που θέλει να μεταφέρει ή να πετύχει το ΕΦΣΙ δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει μια φιλόδοξη ισορροπία μεταξύ προσθετικότητας και απαιτήσεων αφενός και αφετέρου των δυνατοτήτων που προσφέρει παραδείγματος χάρη συμμετοχή περιφερειακών και τοπικών τραπεζών στην ανάπτυξη έργων. Κυρία Τσάνοβα, θέλω να σας ρωτήσω το εξή. Τι εγγυήσεις μπορείτε να μας προσφέρετε για να αποφευθούν να έχουμε κακή επιλογή ή ανεπαρκή έλεγχο έργων και να επομιστούν ε, το τίμημα οι πολίτες ή μπορείτε να δεσμευτείτε ε, ότι στη διαχείρισή σας δεν θα έχουμε ασύμβατες επενδύσεις με τους στόχους της Ευρώπη 2020, η πυρηνική ενέργεια που μένει εκτός ως τομέας και μπήκε ενεργειακή απόδοση στη θέση της κτλ. κτλ. Ή πιο γενικά. Τι θα κάνουμε ώστε το ΕΦΣΥ να μην επιδεινώσει τις ε, αυξηνόμενες ανισότητες μεταξύ διαφόρων περιφερειών. Δηλαδή, με άλλα λόγια, πώς θα πηγηθεί το ΕΦΣΥ να μην είναι απλά ένα νέο χρηματοοικονομικό ή χρηματοδοτικό εργαλείο και να μην ε, απλά δίνει περισσότερο κεφάλαιο στην ΕΤΕΠ. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε με ευφυή βιώσιμο τρόπο τα κονδύλια αυτά προς όφελος όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το βασικό μου ερώτημα. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ο Μπάς Σας ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήσεις έχω σχετικά με τον πίνακα επιδόσεων. Τον αναφέρατε αρκετές φορές, γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω. Καταρχάς, στο παράρτημα αναφέρεται ότι ο πίνακας επιδόσεων θα χρησιμοποιηθεί ως ένα εργαλείο έτσι ώστε η Επιτροπή Επενδύσεων να δημιουργήσει προτεραιότητες. Όμως ο πίνακα επιδόσεων προς το παρόν έχει μια αξιολόγηση για τους διαφορετικούς πυλώνες. Εσείς πώς θα τον χρησιμοποιήσετε έτσι ώστε να ε, αξιολογήσετε τα έργα πραγματικά. Θα ήθελα να μάθω πώς θα το κάνετε αυτό βασισμένοι σε αυτό τον πίνακα επιδόσεων. Έπειτα, συνεχίζοντας, αναφέρεται ότι ο πίνακας επιδόσεων προβλέπει μία ανεξάρτητη αξιολόγηση των εγγύσεων που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς ε, θα ήθελα να μάθω πώς βλέπετε αυτήν την ανεξαρτησία του πίνακα επιδόσεων, πώς εσείς θα ε, πείτε στην Επιτροπή ΕΚΟΝ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πώς ακριβώς χρησιμοποιείται ο πίνακα επιδόσεων για τα διάφορα έργα, πώς εσείς θα αιτιολογήσετε αυτήν την διαφάνεια, πώς θα την εξηγήσετε σε εμά υπό τον εφισταμένο κανονισμό. Κυρία Τσάνοβα, έχετε το λόγο. Βλέπω πως έχετε αποθέσει τις ελπίδες σας σε μένα για να διασφαλίσω ότι όλα θα εφαρμοστούν έτσι όπως πρέπει. Ελπίζω να καταφέρω να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων. Ε, να σας πω βέβαια ότι ο κανονισμός υπάρχει και εγώ απλά δεν θα κάνω τίποτα άλλο από το να τον ακολουθήσω. Τώρα, πώς θα αποφύγουμε την επιλογή λάθος έργων. Πιστεύω προσωπικά ότι πρέπει από νωρίς να ενσκύψουμε πάνω στα έργα αυτά έτσι ώστε να δούμε τι ακριβώς γίνεται, να δούμε πως ε, ό,τι ζητά την υποστήριξη του ένση την αξίζει πραγματικά έτσι όπως προβλέπει ο κανονισμός. Ο πίνακας επιδόσεων θα έχει κάποιους δείκτες που θα αξιολογούν το κάθε έργο ξεχωριστά όταν αυτό θα παρουσιάζεται στην Επιτροπή Επενδύσεων και θα αιτιολογεί λοιπόν το σκεπτικό βάση του οποίου επελέγει το κάθε έργο και προτάθηκε στην Επιτροπή Επενδύσεων για έγκριση. Εγώ προσωπικά θα ζητήσω πληροφορίες για το πώς αιτιολογήθηκα η έγκριση του κάθε έργου και εάν καταφέρουν να πείσουν εμένα και τα υπόλοιπα μέλη της ε, Επιτροπής ότι αξίζουν αυτά τα έργα χρηματοδότηση, τότε θα τα εγκρίνω. Πράγματι, τώρα υπάρχουν τέσσερις πυλώνες στον πίνακα επιδόσεων. Κάθε πυλώνας έχει δείκτες. Το σημαντικό όμως είναι εμείς και εσείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, τοποθετηθούμε ως προς το τι θεωρούμε πως είναι σημαντικό, ποιος πυλώνας είναι σημαντικός. Όταν λοιπόν έχουμε τα έργα και μία βάση δεδομένων για αυτά, θα έχουμε την υποχρέωση να υποβάλουμε εκθέσεις σε εσά εγκαίρως και τακτικά. Και έτσι λοιπόν θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα διαλόγου που θα μπορούμε να σας ενημερώσουμε για την πρόοδο των εργασιών μας και εσείς να δείτε πώς ακριβώς ε, λειτουργούμε και τι ακριβώς γίνεται, αν έχουμε αποτελέσματα. Αυτός λοιπόν ο πίνακας επιδόσεων είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο για την Επιτροπή Επενδύσεων. Τη βοηθά να λάβει αποφάσεις, έχει πληροφορίες τις οποίες έχετε ήδη εκφράσει την επιθυμία να ε, έχετε και δίνει έμφαση σε συγκεκριμένα κριτήρια Προσθετικότητα, κινητοποίηση ιδιωτικού κεφαλαίου για παράδειγμα, τη θέμενη αξία στους ε, ευρωπαϊκούς στόχους πολιτικής κτλ. Ευχαριστούμε πολύ για το ομάδα EFTD, ο Μαρκο Τζάνι. Ναι, ευχαριστώ. Έχω μία ερώτηση κατά την απόψή σας. Ποιος θα είναι ο ρόλος του ΕΦΣΙ Σήμερα στην Ευρώπη, όπως γνωρίζουμε, πολλές επιχειρήσεις δεν επενδύουν όχι γιατί δεν έχουν ρευστότητα ή χρήματα, αλλά γιατί δεν υπάρχει ζήτηση. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα σήμερα στην Ευρώπη, το οποίο... στο οποίο οφείλεται και η έλλειψη επενδύσεων εκ μέρους των επιχειρήσεων. Κατά την άποψή σας, πώς θα δράσει το ΕΦΣΙ ώστε να τονώσει τη ζήτηση περισσότερο από την προσφορά. Δεύτερον, κατά την άποψή σας, ποιοι είναι οι τομείς ε, που μέσω του ΕΦΣΙ θα μπορούσαν να υποστηρίξουν πιο αποτελεσματικά την ζήτηση. Και δεύτερον, ε, πιο γρήγορα σε περίπτωση που επιλεγείτε ως αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του ΕΦΣΙ, πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα που θα υπάρξει με ιδιωτικές επενδύσεις ε, σε τομείς που αφορούν ε, βασικές υπηρεσίες όπου ενίοτε η ιδιωτικοποίηση προκαλεί αποκλεισμό ενός μέρους του πληθυσμού από τέτοιες υπηρεσίες όπως για παράδειγμα η εκπαίδευση. Κούβρι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ γρήγορα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Είναι σημαντικό να εμπλακούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις περισσότερο από ότι μεγάλες. Εσείς ε, συμφωνείτε με αυτή τη δήλωση. Πώς θα διασφαλίσετε ότι θα είναι πολλές ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα έχουν πρόσβαση στο Ταμείο του Γιόνκερ δεδομένου ότι πολλές έχουν αποκλειστεί. Και μετά όσον αφορά τον αξιολόγηση για το ζήτημα που σχετίζεται με το Κάστορ. Ε, κατά την άποψή σα, είναι μια επένδυση που θα μπορούσε να ενταχθεί. Α, ε, συγγνώμη, το Κάστορ, η αποθήκευση φυσικού αερίου θα μπορούσε να ενταχθεί στι επενδύσει ε, του ΕΦΣΥ. Κυρία Τσάνοβα. In terms of, um, Να ξεκινήσω με το πρώτο ερώτημα. Θα διαφωνούσα ελαφρώς ότι η ρευστότητα είναι ένα πρόβλημα. Έχουν δείξει πολλές μελέτες ότι δεν είναι η ρευστότητα το πρόβλημα. Αλλά περισσότερο η αχορταγία των κερδοσκόπων. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι πώς θα ξεκλειδώσουμε την επενδυτική ικανότητα και πώς θα υπάρξει επιμερισμός κινδύνων μεταξύ τραπεζών που είναι πρόθυμες να δανείσουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, αλλά απαιτώντας ταυτόχρονα λιγότερες εγγύσεις γιατί θα υπάρχει εγγύηση του εύση στο πρόγραμμα αυτό, το εκάστοτε έργο δηλαδή. Επίσης θα πρέπει να έχουμε κάποιο κίνδυνο, ρίσκο για να μπορούν να έρθουν και άλλοι από τον ιδιωτικό τομέα για να επενδύσουν στα έργα. Αυτό νομίζω ότι καλύπτει και το ερώτημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πολύ σωστά είπατε ότι στις αναπτυγμένες οικονομίες οι ΜΜΕ παρέχουν τις περισσότερες θέσεις εργασίας στη χώρα. Και από ό,τι έχω δει, τουλάχιστον στα πιο νέα κράτη-μέλη, το πρόβλημα με τις ΜΜΕ είναι ακριβώς η έλλειψη χρηματοδότησης. Γιατί οι τράπεζες πρέπει να πληρώσουν κάποιες απαιτήσει, απαιτούν υπερβολικά μεγάλες εγγύησεις ε, ή δεν μπορούν να δανειστούν ε, τα ποσά ή Ε. Άρα θέλουμε και επιμεσμό κινδύνων και ε, προϊόντα για τις ΜΜΕ και να εστιάσουμε στις ΜΜΕ για να αναπτυχθούν και να συνεχίσουν να παρέχουν περισσότερες θέσεις εργασίας για τους πολίτες των χωρών. Για την αποθήκευση φυσικού αερίου είναι σαφή τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Πρέπει να τηρούνται αυτά τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την επιλογή των έργων που είναι και προσθέμενη αξία δημιουργία θέσεων εργασία, συμβολή στην ενεργειακή απόδοση, στρατηγικέ υποδομέ. Αυτά είναι τα κριτήρια φιλεξιμότητα. Ευχαριστώ. Πρόεδρο για την ομάδα ΙΕΝΕΦ. Κύριο Ζόλτεχ. Μονό. Ουδής. Δύο λεπτά σας απομένουν, κυρία μου, για να συμπληρώσετε και να ολοκληρώσετε. Well, thank you very much for... Ευχαριστώ πολύ που μου αφιέρεσατε χρόνο για να συναμιλήσουμε απόψε. Πρέπει να πω ότι έχω εντυπωσιαστεί από το επίπεδο των συζητήσεων και των ερωτήσεων που θέσατε. Πραγματικά δεν βλέπω την ώρα να πιάσω αυτή τη δουλειά και να συνεργαστώ μαζί σας ε, στο μέλλον ε, και ελπίζω ότι θα συνεργαστούμε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους λοιπούς και ότι σε τρία χρόνια θα μπορούμε να δηλώσουμε με περηφάνεια ότι το FC υπήρξε επιτυχές. Δεν θα είναι εύκολο το εγχείρημα, αλλά είμαι αισιόδοξη. Πιστεύω ότι με την κοινή μας προσπάθεια θα το πετύχουμε. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Έχουμε, έχει ήδη περάσει η ώρα, οπότε να σας αφήσω να πάτε να πιείτε ένα ποτό είναι να Ευχαριστούμε πολύ, αξιότιμη κυρία. Έχουμε ολοκληρώσει τις ακροάσεις. Θα σταματήσουμε τώρα για πέντε λεπτά. Δέκα λεπτά. Και καλό τους υποψήφιους και τους ε, παρατηρητές να εγκαταλείψουν την αίθουσα. Θα επανέλθουν αργότερα γιατί η ψηφοφορία βέβαια είναι δημόσια.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 But Συγγνώμη, από όσο καταλάβα, ε, πολύ σύντομα θα πρέπει να κάνουμε την ανταλλαγή απόψεων, το οποίο είναι μόνο για μέλη. Οπότε τα μη μέλη θα πρέπει να αποχωρήσουν μετά. Αυτή είναι η κανονική διαδικασία. Οπότε να ζητήσω να είναι παρόντα μόνο μέλη και ο εισηγητής να πάρει το λόγο για ένα-δύο λεπτά και μετά να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Ε, παρακαλώ λοιπόν οποιοδήποτε γραμματής ε,